Okay, colleagues, um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε και ευχαριστώ όσους είναι παρόντες εγκαίρως. Αυτούς που είναι πάντα εδώ εγκαίρως και το εκτιμώ αυτό. Προσπαθούσα να δω εάν είναι κάποιος από τους ε, εισηγητές μας σήμερα το πρωί ο κύριο Δίαθ Δεμέρα είναι εδώ. Μου είπαν ότι για οικογενειακού λόγου δεν μπορεί να είναι εδώ. Οπότε είναι εδώ η άλλη συγγήτρια, η κυρία Τάνια Φαγιών. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το πρώτο τμήμα είναι το πρόγραμμα καταχωρημένων ταξιδιωτών που θα το παρουσιάσει η Τάνια. Α, να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Επιτροπή. Α, ωραία. Λοιπόν, μια σύντομη εισαγωγή να σας υπενθυμίσω ότι στις 16 Οκτωβρίου η Επιτροπή παρουσίασε στην Επιτροπή μας την τεχνική μελέτη για τα ευφύη συνορατότητα το κεφάλαιο που αφορούσε το κόστος και τα προτινόμενα συστήματα δεν ήταν διαθέσιμο. Σήμερα λοιπόν, όπως ε, είχαμε πει και τότε, η Επιτροπή θα μας παρουσιάσει αυτή την ανάλυση για το κόστος. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα πάρει το λόγο η συγκίτριά μας κυρία Τάνια Φαγιών και φυσικά όσοι άλλοι θέλουν να πάρουν το λόγο μετά θα έχουν δυνατότητα. Ο κύριος Ρόζενμπεργκ λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, παρακαλώ όχι πάνω από 15 λεπτά και μετά θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι και αν χρειαστεί θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Παρακαλώ κύριε Ρόζενμπεργκ. Κάντε την παρουσίασή σας και μετά θα παρέμβουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα την οικονομική πτυχή του προγράμματος αυτού. Θα το συνδέσω με τα κύρια πορίσματα της έκθεσης που σας υποβλήθηκε ήδη στις 16 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω το πλαίσιο. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για τεφή σύνορα το Φεβρουάριο του 2013 ως αντίδραση στην ανάγκη εξυγχρονισμού της διαχείρισης των σύνορων Σέγγεν 2 στοιχεία, ε, σύστημα εισόδου-εξόδου και σύστημα καταχωρημένων ταξιδιωτών. Κατά την πρώτη τους αντίδραση, οι συνομοθέτες εξέφρασαν ανησυχίες για το κόστος και το τεχνικό τμήμα. Το Φεβρουάριο 2013 έγινε η συμφωνία να εξετάσουμε κατά πόσο συνολικά το πρόγραμμα για να δούμε αν είναι εφικτό. Είχε δύο φάσεις. Πρώτη, η τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο και το οικονομικό τμήμα που υποβλήθηκε τέλος Οκτωβρίου και μετά η φάση δοκιμής, το πιλωτικό όπως λέγεται πρόγραμμα που είναι σε φάση προετοιμασίας και θα εφαρμοστεί τον ερχόμενο Μάρτιο. Όπως είπε χθε ο κύριος ε, Πίτροπος Αβραμόπουλος, μετά τη φάση δοκιμής που περιμένουμε ότι θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο του 2015, όσο το δυνατόν πιο σύντομα η Επιτροπή θα υποβάλει όχι αναθεωρημένη, αλλά μια νέα νομοθετική πρόταση. Τέλη 15 ή αρχές 16. Και παράλληλα οι προτάσεις ε, του 2013 θα αποσυρθούν. Με τις νέες προτάσεις θα ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που εξέφρασε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για να δούμε τώρα την ίδια τη μελέτη που αφορά το κόστος. Κύριος στόχος του κεφαλαίου για το κόστος είναι να έχουμε ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για το πόσο θα μας στοιχήσουν αυτά τα δύο συστήματα του EES και του RTP. Τι θα στοιχεί στην Κομισιόν, τι θα στοιχεί στα κράτη-μέλη. Δεύτερος στόχος ήταν να εκτιμήσουμε εάν ο προπολογισμό για το πρόγραμμα, το πακέτο αυτό, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών 14 ή 20 που είναι 791 εκατομμύρια, θα κάλυπτε το κόστος που είχαμε υπολογίσει. Ο προπολογισμό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι επαρκής για να καλύψει τρία χρόνια ανάπτυξης 17-19 και ένα έτος λειτουργίας αν πάρουμε τι προτάσει του 2013 ω βάση, το κόστο συνολικά θα είναι 430 εκατομμύρια. Και αν κάνουμε μια εκτίμηση με βάση αυτό στην επταετή περίοδο, που συμπίπτει με το πλαίσιο, το δημοσιονομικό είναι τεχνητό αυτό αλλά χρήσιμο, το συνολικό κόστο ανάπτυξη και λειτουργίας ε, προβλέπουμε να είναι 622 εκατομμύρια, 22% περίπου λιγότερο από το προπολογιστέν μέχρι στιγμή κόστος. Γιατί είναι τόσο σημαντική η μείωση. Πολλοί λόγοι, δύο κυρίως. Πρώτος, από τότε που κάναμε τους πρώτους μας υπολογισμούς, λόγω της αύξησης ε, του ανταγωνισμού στην αγορά, του κλάδου αυτού, έχει μειωθεί το κόστος ε, των υπηρεσιών δικτύου. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Δεύτερος, εισαγάγαμε μια νέα, ένα νέο στοιχείο, το λεγόμενο εθνικό ολοκληρωμένο σημείο επαφής. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε επιμέτρο εθνικά συστήματα που να συνδέονται με το κεντρικό σύστημα και με βάση τη μελέτη φαίνεται ότι έχουμε πολύ λιγότερο κόστος και είναι πολύ πιο εφικτό ένα τέτοιο σύστημα. Um, για μία ε, πλατφόρμα διάδρασης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όλα ε, τα κράτη-μέλη. Το 2013 ε, στις προτάσεις της Κομισιόν σκεφτήκαμε δύο συστήματα χωρίς άμεση αλληλεπίδραση και σύμφωνα με τη μελέτη αν υπάρχει ένα σύστημα με EES ε, και RTP ε, λειτουργίες. Αυτό θα είχε πολλές ε, δυνατότητες, θα μπορούσε να καταγράφει τα δεδομένα των ταξιδιωτών με καλύτερο τρόπο και επίσης θα μείωνε και το κόστος οι οικονομίες ενός και μοναδικού συστήματος θα σήμαιναν 49 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα έτη ε, επειδή υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στην ανάπτυξη του δικτύου όπως επίσης και ε, το κόστος συντήρησης κλπ. Αν κανείς κάνει μια παρεκβολή για μια περίοδο 7 ετών, οι οικονομίες θα ήταν περίπου 17 εκατομμύρια. Μιλάμε λοιπόν για σημαντικό ποσό. Είναι σημαντικό να έχουμε καλύτερα ένα ενιαίο σύστημα ε, αντί για περισσότερο. Περισσότερα. Κάτι ακόμη. Η σχέση με το σύστημα ε, θεωρήσεων, το VIS. Ε, κοιτάμε πώς μπορούμε να έχουμε μία σύνδεση μεταξύ του VIS και του νέου συστήματος εφιών συνόρων, να έχουμε το ERS και το RTP από την αρχή της ανάπτυξης κάτι το οποίο θα σήμαινε βέβαια επιπλέον κόστος 39 εκατομμυρίων. Και αυτό οφείλεται στην ανάγκη να αμβλύνουμε τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου συστήματος επί τη βάση ενός υπάρχοντος συστήματος VIS, ε, το οποίο είναι αποτελεσματικό σε 30 χώρες επί καθημερινής βάσεως. Είναι λοιπόν περίπλοκο από τεχνικής απόψεως. Και ε, επίσης οι δοκιμές ε, και η έναρξη ισχύω θα ήταν αρκετά δύσκολη και επομένω δαπανηρή σε σχέση, για να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα που να μπορεί να στέκεται από μόνο του. Η μελέτη επίσης εξηγεί ότι αν έχουμε μια προγροδευτική ε, ε, ολοκλήρωση του ΙΑΡΕΣ και του RTPS ε, χρησιμοποιώντας στοιχεία του VIS από την αρχή του προγραμματισμού και του συστήματος εφιών συνόρων, θα ήταν καλό εντός μερικών ετών να συγχωνευτούν τα δύο συστήματα. Αυτό θα ήταν πολύ ασφαλίστερο. Βέβαια θα ήταν το, το κόστος ανάπτυξης λίγο μεγαλύτερο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια θα εξοικονομούσε κανείς χρήματα. Και έτσι θα υπήρχε στο τέλος, θα υπήρχαν οικονομίες 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το αρχικό ε, σενάριο. Όσον αφορά τώρα τον ε, ταυτοποιητή βα... βα... βιομετρικών στοιχείων. Ε, αναφερθήκαμε στα αποτυπώματα ως ε, τα βασικά βιομετρικά στοιχεία, ε, τέσσερα τελικά αποτυπώματα για το RTP. Επειδή υπάρχει όμως τεχνολογική εξέλιξη στο θέμα των βιομετρικών, η μελέτη αναφέρει επίσης και τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου. Για, πολλά μπορούν να υποθούν για τα υπέρ και τα κατά αυτών των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά από απόψε ως κόστους και μόνο φαίνεται ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα σενάρια είναι σημαντική. Ίσως όχι τόσο μεγάλη όσο θα σκεφτόταν κανείς. Η διαφορά μεταξύ του, της πιθανότητας ε, να έχουμε 8 δακτυλικά αποτυπώματα ε, αντί για 4 είναι λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια τετραετή περίοδο. Το σενάριο που λέει ότι θα χρησιμοποιούμε μόνο αναγνώριση προσώπου και καθόλου αποτυπώματα είναι το φθηνότερο σενάριο, όπως θα φανταζόταν κανείς, 23 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τα 8 αποτυπώματα. Αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση με τα δίκτυα, με το νόγκο των δικτύων, γιατί όσο περισσότερα στοιχεία συλλέγει κανείς, τόσο περισσότερα δεδομένα επεξεργάζεται και τόσο υψηλότερο το κόστος. Τώρα, ε, η πρόσβαση στην επιβολή, της επιβολής του νόμου, των αρχών επιβολής του νόμου. Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει πρόβλεψη τέτοιας πρόσβασης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα έχει θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη ανάγκη αναλογικότητα της πρόσβασης των αρχών επιβολή του νόμου και ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταδειχθεί. Βεβαίως η μελέτη δεν ασχολήθηκε με τις πολιτικές πτυχέ του θέματος, αλλά υπολόγισε βεβαίως το τι θα στήχιζε ε, να ε, υπάρχει πρόσβαση από τις αρχές επιβολής του νόμου και φαίνεται ότι το κόστος υλικού και λογισμικού για την αναζήτηση κάποιων αποτυπωμάτων δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. 2,5 ε, εκατομμύρια ευρώ για συντήρηση, για κόστος λειτουργίας ε, περίπου 1,2 ε, εκατομμύρια Ε, εάν, ε, όλα αυτά εάν η αποθήκευση γίνεται για μια περίοδο 90 ημερών μετά τη στιγμή της εξόδου. Αυτό είναι κάτι που προβλέπεται στο βασικό σενάριο. Αν παραταθεί αυτή η περίοδος κράτησης των δεδομένων σε ένα χρόνο για παράδειγμα, τότε το κόστος αυξάνεται 26 εκατομμύρια ευρώ για μια τέτοια παράτηση, ε, παράταση. 2,3 εκατομμύρια ήταν το αρχικό ποσό που ανέφερα προηγουμένως. Αν γίνει η παράταση σε 5 χρόνια, τότε το κόστος ανάπτυξης θα είναι 32 εκατομμύρια και ετήσια συντήρηση ε, πάνω από 9 εκατομμύρια κατέτος εδώ λοιπόν βλέπουμε το σοβαρό αντίκτυπο και για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη η κατάσταση πρέπει να αναφερθεί ότι η παράταση της ε, προβλεπόμενης ε, περίοδου ε, είναι κατά την άποψη του εισηγητή αλλά και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαραίτητη ε, για την ταχύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων στα σύνορα αλλά και για τους ταξιδιώτες γιατί διαφορετικά οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επανακαταχωρούνται, κάτι το οποίο θα δημιουργούσε μεγαλύτερη παρακόλληση στα σύνορα και πει να το δούμε ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως της πρόσβασης της αρχής ε, των αρχών επιβολής του νόμου. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών, η πρόταση του 2013 είχε συμπεριλάβει ε, το RTP token, ε, το οποίο θα χρησιμοποιούσε το σύστημα. Ένα τέτοιο ε, εργαλείο θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο και το ίδιο θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να χρησιμοποιούμε μια αναγνωρίσιμη ζώνη, αναγνώσιμη ζώνη πάνω στο εισιτήριο. Και αυτό θα σήμαινε εξοικονόμηση 15 εκατομμυρίων για το σύστημα. Η μελέτη επίσης αναφέρει ότι υπάρχει μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό σύστημα που θα μείωνε τους επιπλέον πόρους που θα χρειάζονταν στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των αιτήσεων. Η ιδέα είναι να επιτρέψουμε σε κάποιους που ήδη έχουν καταχωρηθεί στο ΙΕΣ να μπορούν να ζητήσουν ε, καθεστώς άρτη είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ε, ρεαλιστικό μοντέλο και αυτή η επιλογή από απόψεως οικονομικής δεν θα έχει ιδιαίτερο οικονομικό αντίκτυπο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά όπως είπα μπορεί να έχει ένα, εποφελές, ε, ένα αντίκτυπο σε, στους εθνικούς προϋπολογισμούς για τα συστήματα τώρα πληροφορική για τι αεροπορικέ εταιρείε και για του ταξιδιώτε. Επειδή τα διαβατήρια δεν θα σφραγίζονται πλέον στο μέλλον, προτείνει η μελέτη να έχουν οι ταξιδιώτε τη δυνατότητα να λάβουν και να ζητήσουν πληροφορίε για το μέγιστο αριθμό ε, ημερών ε, που του επιτρέπεται να παραμείνουν ε, στη ζώνη Σέγγεν, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα φαίνεται πια ω πληροφορία στο διαβατήριο. Μία παρόμοια λύση θα μπορούσε να υπάρχει και για τι τις αεροπορικές εταιρείες ώστε να μπορούν να επαληθεύουν ε, την ισχύ της θεώρησης ε, και το, το καθεστώς του ταξιδιώτη. Κάτι το οποίο δεν αναφερόταν στην πρόταση του 2013 και δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό οικονομικό σενάριο. Πρέπει να δούμε πώς θα τα οργανώσουμε όλα αυτά στην πράξη. Υπάρχουν ε, πολλές αναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Και είναι σημαντικό και θέλω να το επισημάνω ότι ούτε οι ταξιδιώτες ούτε οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα. Η ουσία είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα σύνολα δεδομένων ε, ε, με απαντήσεις τύπου ναι ή όχι από τον ταξιδιώτη ε, και την αναφορά των ημερών που τους επιτρέπεται να παραμείνουν στη ζώνη Σέγγεν. Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα θα επιζητούν μια ε, επένδυση 4,2 εκατομμυρίων και 1,5 εκατομμυρίου για λειτουργικό κόστος κατέτος. Το κόστος τώρα του πιλωτικού ε, προγράμματος. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει ε, δοκιμή ε, πλήρης του ΙΕΣ e και του RTP. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα είναι το σύστημα. Όμως έχει γίνει μια προσωμείωση προς τα κάτω για να ελέγξουμε κάπως το σύστημα μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του κεντρικού συστήματος. Εθελοντικά τα κράτη-μέλη θα δώσουν κάποιους, κάποιο, παρέχουν κάποιο προσωπικό και έχει υπολογιστεί ότι ο κόστος, το κόστος της δοκιμής ε, σε έξι σημεία διέλευσης των συνόρων ε, ε, σε χερσαία σύνορα θα ανέλθει σε 2,3 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των σημείων διέλευσης ε, θα είναι υψηλότερος όμως στην πραγματικότητα και μπορεί να χρειαστεί επιπλέον, να χρειαστούμε επιπλέον δοκιμές. Είναι κάτι το οποίο είχατε αναφέρει και εσείς ε, στο ε, γράμμα που είχατε αποστείλει στον Επίτροπο πριν από δύο εβδομάδες. Βέβαια όλα αυτά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμπέρασμα. Το νέο σύστημα ευφυών συνόρων, όπως διαμορφώνεται, μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ε, υπάρχοντος προϋπολογισμού του ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Πολλές ακόμη προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. η αρχιτεκτονική του συστήματος, η επιλογή των βιομετρικών στοιχείων, η συλλογή και η διατήρηση των δεδομένων, η επιτάχυνση της διαδικασίας, όλα αυτά σημαίνουν κάποιο κόστος. Αλλά αυτή η μελέτη θα σας δώσει τις ε, λεπτομέρειες και θα δώσει ε, τη δυνατότητα σε όλους αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σωστές επιλογές στην επερχόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόζενμπεργκ. Η κυρία Τάνια Φιόν, ε, η ησυχήτριά μας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα στοιχεία που παρουσίασε σε αυτή τη μελέτη. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω γιατί βρισκόμαστε τη μέτωμη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κυρίως επειδή γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μετά την πολιτική πάση θα αποσύρει αυτή την πρόταση και θα προτείνει μία άλλη, μάλλον θα αναθεωρήσει την ήδη υπάρχουσα. Και δεν γνωρίζουμε ποια στοιχεία θα είναι στην καινούργια στην ουσία. Τώρα συζητάμε τα αποτελέσματα της μελέτης με διάφορες, ε, διάφορα σενάρια που αφορούν το κόστος και τις διάφορες αναλυτικές λύσεις ε, επί των οποίων καλούμε θα να αποφασίσουμε. Λυπάμαι που δεν είναι ο συνάδελφος Μέρα εδώ με τον οποίο είχαμε συζητήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μεταξύ μας. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο ξέρουμε τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που θέτουν τα στοιχεία που παρουσιάζεται. Εξακολουθώ να τρέφω τον ίδιο φόβο. Το βασικό ε, ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ακόμα και μετά την σύνταξη αυτής της μελέτης Πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν κατάφερε να αποδείξει ότι αυτά τα συστήματα είναι πραγματικά αναγκαία και ότι θα ε, καταλήξουν σε μια προστιθέμενη αξία. Στόχος μας είναι η ασφάλεια από τη μία πλευρά και διευκόλυνση των ταξιδιωτών από την άλλη. Και το κόστος το οποίο αναφέρεται να εξαρτάται από τις διάφορες εκδοχές, τα διάφορα σενάρια που θα επιλέξουμε στο μέλλον. Συνεχίζω να πιστεύω ότι το βασικό μέλημα του Κοινοβουλίου θα είναι η πρόσβαση σε ό,τι αφορά το θέμα της δίωξης. Εδώ μιλάμε για, το, για τις υπηρεσίες δίωξης, το κόστος όμως είναι υψηλότερο. Το βασικό μας μέλημα είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε κάτι τέτοιο και δεν προβλεπόταν στην αρχική νομοθεσία. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με την Ιταλική Προεδρία. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι οι χώρες μέλη είναι σαφώς υπέρ του να υπάρχει πρόσβαση των διοκτικών αρχών και η Επιτροπή είπε ότι δεν είναι αυτή τη άποψη. Είναι δύσκολο λοιπόν να συζητήσουμε αυτό που θα περιέχεται στη νέα πρόταση. Είναι όμως κάτι που μας προβληματίζει και ε, η πρόσβαση των ιδιοκτικών αρχών συνεπάγεται πρόσωπο προσώρο 60 εκατομμυρίων ευρώ. Εξαρτάται αν θα καλύψουμε ένα διάστημα 5 ετών. Τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε 70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κάτι που θα απαιτήσει μια εντελεχή πολιτική συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Έχουμε μια μελέτη, έχουμε μια πιλωτική φάση η οποία θα εφαρμοστεί, θα ξεκινήσει του χρόνου ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε. Από την άλλη πλευρά, η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι οι χώρες μέλη πρακτικά εφαρμόζουν αυτούς τους μηχανισμούς και την τεχνολογία παρόλο που η τελική νομοθεσία, η συμφωνία δεν έχει περατωθεί ακόμα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την επικάλυψη, το κόστος του συστήματος. Νομίζω λοιπόν ότι παραμένει το βασικό ερώτημα, δηλαδή τι θέλουμε να επιτύχουμε, ποιος είναι ο στόχος μας και αυτό βρίσκεται σε κάποια ισορροπία με το κόστος και την πρόσβαση των διοκτικών αρχών. Δεν θα ήθελα να έρθω σε λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκέντρωση δεδομένων και το ποια θα είναι τα δεδομένα αυτά κτλ. Το άλλο που θα επιθυμούσα ε, να γνωρίζω από την Επιτροπή είναι πώς θα μπορούσατε να αιτιολογήσετε ότι για το συστημα καταχώρηση καταχώρησης εισόδου-εξόδου θα αφορά και τους ε, πολίτες μιας χώρας. Το κόστος θα είναι λιγότερο κατά 300 εκατομμύρια από ότι ε, το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών που αφορά 9 εκατομμύρια επιβάτες. Πού φύλλεται αυτή η διαφορά, γιατί το σύστημα αυτό είναι τόσο περισσότερο ακριβό. Θα επιθυμούσα να έχω μια απάντηση. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι ζητήσαμε στην επιστολή μας πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ε, αρμόδιο επίτροπο. χθε ε, είχαμε μια συζήτηση για τα smart borders. Ε, ζητήσαμε να γίνει μια διμερή συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων, δηλαδή τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Έχουμε διαφορετικές πληροφορίες Έχουμε πολλές απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα έτσι ώστε να στα συζητήσουμε στην Επιτροπή και μετά να ενημερώσουμε αντιστοίχω τις χώρες μας. Ε, η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη και πραγματικά να τι θα κάνουμε εάν δεν συνεργαστούμε, αν δεν εργαστούμε εκ παραλίλου. Ευχαριστώ πολύ για την πελέτη, ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες και ελπίζω να υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίε από τη δική σα πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα μιλήσουν τα μέλη και μετά θα περάσουμε στην Επιτροπή ο κύριος ε, Κάλλου, κάποιο άλλο μέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω αυτή τη σημαντική μείωση του κόστου ε, του smart borders ε, σε σχέση με την αρχική πρόταση του 2013. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η μείωση επετεύχθη χωρίς να υπάρχει επίπτωση επί της ποιότητας. Αντίθετα, ε, υπήρξε βελτίωση της ποιότητας και αφαιρώντας στοιχεία που δεν χρειάζονται, όπως για παράδειγμα ένα ξεχωριστό πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών. Όταν συζητάμε θέματα που αφορούν το κόστος θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το να μην έχουμε ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα στα εξωτερικά συστήματα συνεπάγεται πιο μακριές ε, ε, ουρές ε, αναμονής και περισσότερα λάθη. Από την άποψη ενός κράτου μέρους, η δημιουργία και η συντήρηση ενός τέτοιου συστήματος, είτε καταχώρηση εισόδου-εξόδου, είτε καταχώρηση ταξιδιωτών, είναι επίσης δαπανηρό. Ενώ ε, η αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένη όταν δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Στόχος του πακέτου αυτού είναι να διευκολύνει την διέλευση των συνόρων στους επιβάτες και να μπορέσει το προσωπικό να εστιαστεί στις περιπτώσεις που απαιτούν περισσότερη προσοχή. Επίσης θα μας ε, ε, δώσει πρόσβαση σε χρήσιμε πληροφορίε σχετικά με τα τεκτενόμενα στην περιοχή του Σέγγε, συμπεριλαμβάνοντα και τον αριθμό των ατόμων θα παραμείνουν η πρόσβαση των διοκτικών αρχών θα είναι μια πολιτική άποψη. Όταν όμω κοιτάξουμε το διάστημα διατήρησης των δεδομένων και το κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούνται δακτυλικά αποτυπώματα, ενδεχομένως θα χρειαστεί να κρατήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Όπως είπε όμω, η Επιτροπή, η, ε, ε, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων έχει άλλε επιπτώσει. Το πακέτο Smart Borders θα πρέπει να θεωρηθεί μια μακροχρόνια επένδυση σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλεια Το, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων είναι προ, προαπαιτούμενο για την εσωτερική διακίνηση. Κοιτάζοντα εκ των υστέρων τα πράγματα, ενδεχομένω έπρεπε το σύστημα καταχώρηση εισόδου-εξόδου θα έπρεπε να υπάρχει πριν δημιουργηθεί η ζώνη Σέγγεν. Θα πρέπει τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά δεν θα πρέπει να καταφύγουμε σε υπερβολές. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ένωση ήδη συγκεντρώνει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών ε, δεδομένων σε συστήματα όπως το Eurodact και το τα συστήματα που υφίστανται δεν είναι καινούρια και δεν υπάρχουν δυσεπίλητα προβλήματα. Η αρχή της αναλογικότητας, η ιερή αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ κύριο Βάιο. Η κυρία Βάιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έλεγα. Εμείς οι πράσινοι εκτιμούμε το ότι αποσύρθηκε η πρόταση. Εκτιμούμε επίσης το γεγονό ότι η Επιτροπή δεν έχει την ίδια άποψη με τα κράτη-μέλη όσον αφορά την πρόσβαση των διοκτικών αρχών της αστυνομίας στα στοιχεία αυτά για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Γιατί αυτό δεν είναι αρμοδιότητά της. Τώρα το κόστος Είναι δύσκολο να δούμε αν θα μειωθεί επαρκώς το κόστος. Θέλουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή είναι το εξή. Η Επιτροπή θα ε, τηρήσει αυτά που είπε ότι δεν θα υποστηρίξει τις προτάσεις των κρατών μελών για την πρόσβαση των ε, διοκτικών αρχών στα στοιχεία. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Λέει ο Πρόεδρος. Όχι. Ωραία. Πρώτα την Προεδρία λοιπόν θέλω να ρωτήσω και μετά να συνοψίσει η Κομισιόν και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, σύντομα η Προεδρία και μετά θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τις ερωτήσεις των μελών. Ο κύριος ε, Μενιτσέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Η Προεδρία από την αρχή της εντολής, της θητεία της, ε, θεώρησε το πακέτο Smart Border ως βασική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, η Ιταλική Προεδρία χαίρεται ιδιαίτερα που μπορεί να αναγνωρίσει το έργο όλων των φορέων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτού του ε, φακέλου που έχει ορισμένες πολύπτωκες πτυχές. Σε μια προσπάθεια να θεωρηθεί αυτό το πακέτο των Smart Borders, η ευφυών συνόρων, η Επιτροπή εργάστηκε σκληρά, βάζοντα την ημερησία διάταξη των διαφόρων συνεδριάσεων και των αρμόδιων ομάδων εργασίας το θέμα των ευφυών συνόρων έτσι ώστε να επιτραπεί στην Επιτροπή να προετοιμάσει εντός του τέλους του χρόνου τα ε, δεδομένα που είναι απαραίτητα για να περάσουμε στη φάση των δοκιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους τελευταίους στόχους της Προεδρίας θα είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία από πλευράς ε, ε, του Κορεπέρ σε ό,τι αφορά τις ε, βασικές γραμμές που θα μας επιτρέψουν πώς αυτή η δοκιμαστική φάση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και πώς θα πρέπει να διεξαχθεί. Βεβαίω, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, η Ιταλική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι η όλη άσκηση που αφορά το πακέτο αθειών συνόρων θα έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία από τη στιγμή που θα παράσχει και στους δύο συνομοθέτες ένα φάσμα ε, λύσεων και ε, επιλογών που αφορούν και τεχνικές πτυχές αλλά και την πτυχή που αφορά το κόστος και το όφελος. Βεβαίως τα αποτελέσματα της μελέτης, ε, της δοκιμαστικής ε, φάσης θα αποτελέσουν ένα σημαντικό στοιχείο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις για το πακέτο εφιών συνόρων έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα αφορά και το σύστημα εισόδου-εξόδου, αλλά και το σύστημα ε, και το πρόγραμμα καταχωρήσης ταξιδιωτών. Βεβαίως, στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή τη δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, Μίλησα για την ανάγκη να παράσχουμε και στους δύο νομοθέτες ένα φάσμα δυνατών και πιθανών λύσεων, η Ιταλική Προεδρία είναι απόλυτα πεπισμένη ως προς την ανάγκη συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως θύμισε εξάλλου και ο εισηγητής Φαγιών. Για τον σκόπο αυτό συναντήθηκε πρόσφατα με τους δύο εισηγητές, στους οποίους από τη μία πλευρά παρέθεσε όλες τις φάσεις, όλες τις ψυχέ που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ε, κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Στην, ε, με την ίδια ευκαιρία η Προεδρία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή για να παραθέσει στους δύο εισηγητές Ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε στην επιστολή που στείλατε στον Επίτροπο Αβραμόπουλο και στον Πρέσβη σανίνο στι 28 Εντεκάτου ω προ την ανάγκη στενής συνεργασίας ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Ιταλική Προεδρία λοιπόν βεβαίωσε ότι ελήφθησαν σοβαρά υπόψη αυτά και αυτές οι επιθυμίες που εκφράστηκαν θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών γραμμών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Στην ίδια επιστολή, κύριε Πρόεδρε, εκφράσατε την επιθυμία να υπάρξει μια τριμερής πολιτική συνάντηση ενδεχομένως στις 9 ή 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα. Χθες μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η περίοδος ε, αυτή είναι μάλλον ε, πυρετόδης ε, γιατί είμαστε εν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τι συγκεκριμένε αυτέ οι ημερομηνίες φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο να τα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τον δέοντα ε, πολιτικό συνομιλητή για αυτή τη συνάντηση. Επειδή εμείς ως Προεδρία συνδέσαμε τις εργασίες μας κατά τη διάρκεια όλης, ε, όλου του εξάμεινου της Ιταλικής Προεδρίας με την ε, επερχόμενη Προεδρία της Λετωνίας αναρωτιέμαι μια σκέψη εκφράζω ως προσπάθεια να βελτιώσω το ενδεχόμενο να φύσω το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ των τριών βασικών φορέων, αν θα ήταν σκόπιμο να αναβάλουμε για τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου την ε, τριμερή αυτή συνάντηση με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε από κοινού να ορίσουμε μια ημερομηνία για τη συνάντηση αυτή που είναι καθοριστική σε σημασία για να μπορέσει να επιτευχθεί όλο το πακέτο των ε, ευθειών συνόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την αναλυτική πληροφόρηση που μας δώσατε. Κύριε Ρόζεμπεργκ, θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις της εισηγήτριας και των μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Η βασική ερώτηση είναι αυτή που έθεσε η κυρία Φαγιόν. Είναι αναγκαία αυτά τα συστήματα. Βέβαια η μελέτη δεν απαντάει σε αυτή την ερώτηση. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Κατά την ε, γνώμη της Κομισιόν και αυτό ήταν η βάση και των προηγουμένων προτάσεων. Κατά τη γνώμη λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτω απαραίτητο. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα. Αν δούμε πόσο κόσμο περνάει τα σύνορα και πόσο έχει αυξηθεί η κινητικότητα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα τρέχοντα συστήματα δεν λειτουργούν αρκετά καλά και δεν είναι και αποτελεσματικά από πλευρά κόστου. Γι' αυτό 13 κράτη-μέλη έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία εθνικά συστήματα Έχετε υπόψη στα τα νούμερα. Κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια σφραγίδες μπαίνουν σε διαβατήρια από Ευρωπαίους μεθοριακούς φύλακες. Και αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Δεν μας επιτρέπει αυτο, αυτοματοποιημένο υπολογισμό του πόσοι μένουν παραπάνω. Ούτε μας επιτρέπουν να ταυτοποιήσουμε τα άτομα αυτά. Αυτά ακούμε από όλα τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η απέτηση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι αυτό το νέο σύστημα, αλλά φυσικά με τις βελτιώσεις που συζητάμε. Τα ευφυή e e σύνορα πρέπει να είναι ευφυή. E Γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια να αποτιμήσουμε ε, τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος. Κάνοντας αυτή την μελέτη Αποδεχόμεθα ότι ναι, δεν ήταν ευφυείς οι προτάσεις μας του 2013, αλλά ίσως ε, χρειάζονται ευφυέστερες. Και είναι εφικτό να έχουμε ευφυέστερες προτάσεις. Τώρα, συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί το σύστημα RTP ε, δεν, είναι, δεν είναι ίδια με αυτά που έχουμε στο NIS. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια σύγχυση, το ομολογώ. Αλλά αν δείτε τώρα τις λεπτομέρειες των πινάκων και των στοιχείων θα δείτε τα εξή. Ένα σημαντικό τμήμα του κόστους είναι κοινό και στα δύο συστήματα. Αλλά για λόγους ε, δημοσιονομικής παρουσίασης ε, αποφασίσαμε να τα κατανείμουμε σε δύο ίσα τμήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει μισή χρηματοδότηση σε κάθε σύστημα, αλλά επειδή υπάρχουν ε, κοινά στοιχεία του ενωσιακού με τα εθνικά συστήματα, γι' αυτό τα παρουσιάζουμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν εφαρμοστεί το RTP θα μειωθεί το κόστος στο μισό. Αντίθετα, ολόκληρο το κόστος θα πάει στο εθνικό σύστημα. Αν δούμε τώρα το κεντρικό κόστος του EES και του RTP, το EES κεντρικά θα κοστίσει 94 εκατομμύρια και το RTP 73. Λιγότερο. Αλλά αν τα ε, βάλουμε και τα δύο μαζί κεντρικά, το κόστος γίνεται 130. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα ενοποιημένο κοινό σύστημα, το συμπληρωματικό κόστος του RTP θα είναι 130 94 περίπου 35 εκατομμύρια σε κεντρικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, επειδή είναι λίγο τεχνητή αυτή η παρουσίαση, πρέπει να κάνουμε νέους υπολογισμούς, εάν τελικά δεν συνδεθεί το κεντρικό με τα εθνικά συστήματα. Είναι περίπλοκο. Και φυσικά να συνεχίσουμε τις συζητήσεις επ' αυτού σε τεχνικό επίπεδο. Έγιναν ερωτήσεις για την πρόσβαση των διοκτικών αρχών στα στοιχεία. Συγγνώμη που δεν ε, θα συζητήσω λεπτομέρειες από αυτού τώρα. Ενώπιόν μας έχουμε μια τεχνική μελέτη που δεν εξετάζει την ουσία του ζητήματος. Είναι απλώς τεχνική η προσέγγιση. Όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει αλλάξει. Βεβαίως, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα. Συγγνώμη, πρέπει να υπάρξει ε, απόδειξη ότι είναι σκόπιμη και αναγκαία η προσέγγιση των διοκτικών αρχών επί του RTP και του ES. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό, εσείς. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Δεν έχει αποφασιστεί. Αλλά τέτοιου τύπου θέματα είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να συζητηθούν στον πολιτικό τριμερή διάλογο που προτείνεται ο Επιτροπός μου. Θα σας απαντήσει γραπτός ε, τις επόμενες μέρες. Στην επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρός σας δηλαδή. Ίσως λοιπόν η επιστολή αυτή να αναφέρει ότι τα θέματα που τίθενται θα μπορούσαν να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο ήδη ε, πριν το τέλος του χρόνου ή τον ερχόμενο Ιανουάριο και οπωσδήποτε πριν υποβάλουμε τη νέα μας πρόταση τέλος του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Τάνια, θέλεις να πεις τίποτα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ συναδελφοί για τη συζήτηση που κάναμε. Οι συγγήτρια και οι σκιώδης ε, θα συνανοηθούν για την επόμενη φάση και θα μας πούνε ποια θα είναι. Το επόμενο θέμα, τα εθνικά προγράμματα για τα ταμεία εσωτερικών υποθέσεων. Δεν είναι παρόντες οι συνάδελφοι, οπότε θα κάνουμε μια διακοπή μέχρι τις 10.30. Παρακαλώ να επανέλθετε στις 10.30. Θα σας έλεγα να καθίσουμε και να, και να περάσουμε στα επόμενα σημεία τη ημερησία διαταξή. Ευχαριστώ σου ήρθαν έγκαιρα. Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσουμε σε δύο λεπτά. for patience Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την υπομονή σας, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ήρθαν στην ώρα τους. Δεν έχουμε Σημείο 18. Εθνικά προγράμματα για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην προηγούμενη συνάντηση συζητήσατε τα οικονομικά προγράμματα και σήμερα θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή για να μας μιλήσει για τα εθνικά αυτά προγράμματα. Θα ακούσουμε το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα ως προς τον προγραμματισμό για κάθε χώρα μέλος. Η Επιτροπή μας απέστειλε ορισμένα έγγραφα που έχετε θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και μετά θα μπορέσουμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις από πλευράς των μελών. Παρακαλώ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Σας επισκεφτήκαμε τρεις φορές τις τελευταίες ε, μέρες για να σας εξηγήσουμε ορισμένα θέματα. Ξέρω ότι πολλά από τα μέλη γνωρίζουν το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο Ταμείο. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι παρενθερές με το, ΕΣΥΦΑ, με το Ταμείο ΕΣΕΦ. Το πρώτο βήμα στην αρχή της διαδικασίας αφορούσε τη διεξαγωγή του διαλόγου που έλαβε χώρα πριν από ένα μήνες, ένα χρόνο. Αυτός ο διάλογος ερμήνευσε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στις νομικές, στην οριζόντια στον οριζόντιο κανονισμό. Ο διάλογος με τις χώρες μέλη θα έπρεπε να εξασφαλίσει ότι αυτές οι, πολιτικές είναι φτιαγμένες είναι εξατομικευμένες για κάθε χώρα μέλος μετά από αυτό. Διεξήχθησαν ε, συζητήσεις στην Επιτροπή αυτή σχετικά με το αποτέλεσμα των διαλόγων. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι έχουμε εθνικά προγράμματα που ερμηνεύουν αυτές τις προτεραιότητες, τις εντάσσουν σε εθνικά προγράμματα, έτσι ώστε οι επιλογές αυτές θα αντικατοπτρίζονται στα εθνικά προγράμματα και δεν αποτελούν μια παρέκκληση. Σε ό,τι αφορά θέματα χρονικά, χρονικού πλαισίου, σε κάθε εθνικό πρόγραμμα μπορούμε να πούμε ότι θα χρειαστούν 6 έως 9 μήνες. Αυτές βεβαίως, αυτοί είναι οι υπολογισμοί, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό θα ισχύει για όλα τα προγράμματα. 6 ως 9 μήνες θα απαιτηθούν Όσες χώρες ε, μέλη αρχίζουν να υποβάλλουν, θυμηθείτε ότι οι νομικές πράξεις υπευλήθησαν τον Ιούλιο. Τα πρώτα εθνικά προγράμματα προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σλοβανία, το Ελλαδία, Βέλγιο, Γαλλία και ε, Σλοβακία, Λιθουανία, Ρουμανία, Αυστρία κτλ. Οι χώρες θα έλεγα ότι η υιοθέτηση θα μπορούσε να γίνει τον Απρίλιο του χρόνου. Οι χώρες μέλη που υπέβαλαν αργότερα, όπως για παράδειγμα η Ιταλία που υπέβαλε αυτή τη βδομάδα, η Ισπανία την προηγούμενη βδομάδα, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Πορτογαλία, μερικές από αυτές, για αυτές τις χώρε μέλη η υιοθέτηση των προγραμμάτων θα γίνει τον Ιούλιο-Ιούλιο του 2015. Τώρα, το πώς λειτουργεί αυτό. Οι χώρε μέλη, όπως σας είπα, παίρνουν τα αποτελέσματα των διαλόγων και τα εντάσσουν στα προγράμματα. Μετά ξεκινάει μια διαδικασία, μας τα αποστέλουν, ε, διατυπώνουμε παρατηρήσεις και τις αποστέλουμε σε αυτούς. Βεβαίως, ε, κάθε φορά οι παρατηρήσεις που γίνονται όλο και λιγότερες και οριμάζει όλο και περισσότερο το εθνικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται τρεις ή πέντε φορές έτσι ώστε να πλάσει σε απόλυτη οριμότητα το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι επιτυχάνονται ελάχιστα πρότυπα τα οποία κατά την άποψη της Επιτροπής περιμέ, πε, ε, επιτρέπουν το πέρασμα στην επόμενη φάση. Γίνεται διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους διάφορους φορείς για να υπάρχει βεβαιότητα ότι εξασφαλίζονται πέρα στοιχεία. ό,τι αφορά την ένταξη και την μετανάστευση, θέλουμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι αυτή η συμπληρωματικότητα των ταμείων στον τομέα της προπαρασκευής για πρόσβαση στην αγορά εργασίας υπάρχει. Αυτό ε, σημαίνει ότι μόλις φτάσει, ε, φτάσουν τα πρόβλημα αυτά στο επίπεδο ε, ρημότητας θα μπορούν να εφαρμοστούν. Όπως σας είπα, είμαστε σε φάση προετοιμασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό στην αρχή της επόμενης χρονιάς μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουλίου του 2015 να έχουμε περατώσει την ανταλλαγή αυτή απόψεων γιατί τότε θα έχουμε περισσότερες, περισσότερο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν τη διεξαγωγή ενός εκτενέστερου διαλόγου. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουν φτάσει στο επίπεδο ορίμασης. Ε, να, να θυμίσω ε, ε, ε, βελγικό Ταμείο Ασφαλείας, Γερμανικό, Βελγικό Ταμείο Μετανάστευσης και Ταμείο Μετανάστευσης Λουξεμβούργου. Θα μπορούσα να σας πω ότι στο τέλος της χρονιάς μέχρι 10 εθνικά προγράμματα θα έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο οριμότητα. 10 με 15 μεταξύ του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Μετά θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλο Μαρτίου θα έχουμε φτάσει στα 15 προγράμματα που είναι έτοιμα προ υιοθέτηση και έπονται τα υπόλοιπα Φεβρουάριο, Μάρτιο, μέχρι τον Ιούλιο. Από αυτά τα 5 προγράμματα το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Γερμανία ήδη έχουν ένα προηγμένο σύστημα ε, επανόδου ε, και μετανάστευσης. Θα γίνουν προσπάθειες να βελτιωθούν οι διαδικασίες ασύλου, να γίνουν συντομότερες και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα στάντας των διαδικασιών. Το δεύτερο θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλες ε, οι συνθήκες υποδοχής και οι δυνατότητες υποδοχής και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Βεβαίως θα υπάρχουν και ορισμένες διαφορές. Θα έλεγα ότι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο σε τις ομάδες και τους ε, ασυνόδευτους ε, ανήλικους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας. Χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για να γίνεται μια διαρκής αξιολόγηση και για να μην γίνεται κατάχρηση αυτών των διαδικασιών και βεβαίως ε, θα πρέπει να επιτευχθεί ένα αναγκαίο επίπεδο. Αυτό βεβαίως είναι μια ιδιαιτερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο εστιάζεται περισσότερο σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες και στη σύγκριση της διαδικασίας. Ξέρετε ότι η διαδικασία της άλλες χώρες ε, ήταν έξι μήνες, σαφώς έξι μήνες, γιατί υπέστησαν πίεση στο παρελθόν. Εμείς βραχύνουμε αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιούμε τα κονδύλια ε, για να ε, είναι πιο σύντομες αυτές οι διαδικασίες. Τώρα σε ό,τι αφορά την ένταξη που είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος θα διαπιστώσετε εδώ ότι υπάρχουν διαφορές. Το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο επικεντρώνονται στα μέτρα πρώτης αναχώρησης να ενημερώνονται, να γνωρίζουν πώς είναι η κοινωνία υποδοχής, πώς θα είναι η ένταξη σε διάφορες κοινότητες και αυτό είναι μια συνέχεια, ένα συνεχές από την ε, υποβολή της έντας με τη διεθνή προστασία, αυτό αφορά το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζεται περισσότερο το τι συμβαίνει σε επίπεδο τοπικό, ποια είναι η στάση του πληθυσμού. Οι υπεύθυνοι αναγνώρισαν ότι η στάση των, της Βρετανικής κοινότητας δεν είναι τόσο αρνητική σε ό,τι αφορά τους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες προσπαθούν να κινηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να αναπτύξουν αυτές τις δράσεις και να ενδυναμώσουν τις κοινότητες των μεταναστών. Βεβαίως να υπάρξουν μαθήματα γλώσσας, βεβαίως να υπάρχει επαγγελματική κατάσταση και ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Καταβάλλεται λοιπόν μια προσπάθεια όλα αυτά να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Από την άλλη πλευρά, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θα ε, καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει ένα γενικό πακέτο που θα αφορά την υποδοχή, την ε, ένταξη και τα μέτα πριν από την αναχώρηση για τους δυνητικούς μετανάστες. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή, νομίζω ότι θα πρέπει να σας αναφέρω ότι τα καταφέραμε να πείσουν ορισμένες χώρες να εστιαστούν στην εθελούσια, ε, ε, στον εθελούσιο επαναπατρισμό. Παρόλα αυτά υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή τονίστηκε ιδιαίτερα ο επαναπατρισμός, η επιστροφή γενικά. Τα περισσότερα οικονομικά μέσα του οικονομικού προγράμματος εστιάζονται στην επιστροφή και επιτυχαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, η εθελοντική, εθελουσία επιστροφή, μία ε, ε, επιβεβλημένη ε, επιστροφή για τέσσερις εθελούσιες, Βεβαίω χρησιμοποιούν τα, τα, τα κονδύλια του Ταμείου. Θα ήθελα όμως να αποτίσω φόρο τιμή στην προηγούμενη Επιτροπή. Όταν προτάθηκε ένα ελάχιστο ποσοστό στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Αυτό εξασφάλισε μια ισορροπία στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, επενδύει τουλάχιστον 20% για ε, θέματα ολοκλήρωσης και υποδοχής. Σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν την αστυνομία, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας Βεβαίως τα προγράμματα αφορούν, ε, είναι διαφορετικά, το ένα 30.000, το άλλο 140.000. Ε, Εστιάζουν την προσοχή σε τρία θέματα. Κατάρτιση αξιωματικών της αστυνομίας, οι υποδομές ε, και εξοπλισμός για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις διοκτικές και αστυνομικέ αρχές έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές ε, να είναι ασφαλείς, να γίνονται σεβαστά τα βασικά πρότυπα και να είναι αποτελεσματικά. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία ε, σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα και τις θεωρήσεις, το Eurosur στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια παρέκκληση από το ελάχιστο ποσοστό στην περίπτωση του Βελγίου. Θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Στην περίπτωση του Βελγίου θα χρησιμοποιηθούν τα εγχώρια μέσα έτσι ώστε ε, να διατηρηθούν ε, τα εθνικά πρότυπα. Βεβαίως υπάρχουν περιορισμένα εξωτερικά σύνορα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης αυτού του συστήματος σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχουν προξενία. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν εκεί τα προξενία και μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους και να υπάρχουν και εθνικά κέντρα συντονισμού έτσι ώστε όλες οι αρχές να μπορέσουν να συνεργαστούν με ένα συντονισμένο τρόπο ε, κατά την ε, εποπτεία των συνόρων. Επίσης θα πρέπει να έχουν την ε, βεβαιότητα ότι ό,τι αφορά την διέλευση των σύνορων και τις θεωρήσεις διεξάγεται με έναν ομαλό τρόπο. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά στατιστικά δεδομένα. Είμαστε σε πρώιμη φάση. Αυτό που σας λέω δεν είναι αποτέλεσμα μιας εντελεχού στατιστικής ανάλυσης. Μπορώ όμω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τρει χώρες μέλη, γίνονται σεβαστά τα ελάχιστα ποσοστά. Ε, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η ε, Λετωνία είναι οι αυτέ χώρε, χώρες υπέχουν υποβάλει προγράμματα με ποσοστά που δεν ε, λαμβάνουν υπόψη τους, δεν σέβονται αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να ασκούνται πιέσεις για το σεβασμό των ελάχιστων προσωπών και στο τέλος διαδικασίας ε, εξέτασης οι χώρες αυτές ε, μέλη ή θα πρέπει να τα έχουν σεβαστεί αυτά ή θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν εξηγήσεις. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα και τις θεωρήσεις, Νομίζω ότι έχουμε μια άλλη εικόνα. Επτά κράτη-μέλη δεν τα σέβονται. Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο... Α, Συγγνώμη, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και κάτω χώρες. Αυτές οι χώρες, δεν χρειάζεται βέβαια να τα γράψετε όλα αυτά, μπορώ να σας ε, δώσω τις σχετικές πληροφορίες. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Αυστρία είναι στο ίδιο επίπεδο με το, με το Βέλγιο και τη Δανία, γιατί σε μερικές χώρες είναι πολύ ανεπτυγμένο το σύστημα και πολύ στέρεο, πρέπει απλώς να το διατηρήσουμε και να ε, δεσμεύσουμε δεσμευτούμε στην ενίσχυσή του σε εθνικό επίπεδο, ενώ η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, για παράδειγμα, πρέπει να επιμείνουμε πολύ περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα εθνικά προγράμματα, αν ζητήσουν παρέκκληση, πρέπει να υπάρχει μια καλή αιτιολόγηση και δεύτερον να εξασφαλίσουμε ότι με τα εθνικά τους μέσα μπορούν να να συμπληρώσουν ε, τα ελάχιστα ε, ποσοστά που χρειάζονται. Και να ολοκληρώσω με κάτι ακόμη, δεδομένα για το τομέα του ασύλου, σε γενικές γραμμές ε, επενδύσεις από 20 έως 25% της χρηματοδότησης, η Μάλτα επενδύει 15% στο ε, άσυλο όσον αφορά την ενσωμάτωση 40% και για ε, την ε, επιστροφή Ηνωμένο Βασίλειο και Βουλγαρία είναι οι χώρες που έχουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Um, thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκασόλα. Ένα σχόλιο να κάνω. Ο προκάτοχός μου σας είχε ε, αποστείλει μία επιστολή και εγώ έγραψα σε εσά στην αρχή της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Μιλάτε για τα κράτη-μέλη, δίνετε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα και υποθέτω ότι τα, ε, ε οι συνάδελφοι το ίδιο θα ήθελαν, μία κατανομή λεπτομερή στο σημείωμά σας. Ε, αυτό που μας δώσατε είναι μία αρχή, αλλά ειδικότερα σε σχέση με τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων πρέπει να υπάρχει αναλυτική κατανομή κράτος μέλος του πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια και σε κάθε πρόγραμμα. Και όσον αφορά συγκεκριμένα τα ταμεία αυτά ιστορικών υποθέσεων δεδομένης της ευαισθησίας, ε, ε, την εφελώδη, ε, τον εφελώδη χαρακτήρα των ταμείων αυτών, ε, άσυλο, ε, επανεγκατάσταση κλπ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ πιο πρακτική Καλό είναι λοιπόν το σημείο σας ως αφετηρία, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο σας ζήτησα. Και ίσως μέχρι την αρχή του επόμενου έτους, μήπως θα μπορούσατε όλα αυτά που μας είπατε να τα ε, κατανείμετε λίγο καλύτερα ανακράτος μέλος. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα ενδιαφέρονταν γι' αυτό και θα ήταν και χρήσιμο. Δεν ξέρω αν ε, θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι. Να δώσω τώρα το λόγο για στους συναδέλφους να δω κατά πόσο συμφωνούν με αυτό που λέω. Κυρία Σίπελ πρώτα και μετά η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν αναφερθεί ήδη κάποια από τα θέματα που θα ήθελα να θέσω ε, από τον Πρόεδρο. Αυτά τα εθνικά προγράμματα εγώ δεν τα έχω δει. Θα ήθελα να ακούσω πραγματικά τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Όμως, έχω λάβει γνώση κάποια, κάποιων πραγμάτων για τις προτεραιότητες και για όλους τους ε, διαφορετικούς τομείς τους οποίους χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη τα ε, μία αυτά αλλά ποια είναι τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα συγκεκριμένα μέσα, μέτρα στα κράτη-μέλη και πώς θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτήν την επισκόπηση για να ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάτι ακόμη. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα ταμεία αυτά για επιπρόσθετα μέτρα ή συνεχίζουν ήδη δρομολογηθέντα προγράμματα αλλά δεν τα χρηματοδοτούν πλέον με το δικό τους εθνικό προϋπολογισμό, παίρνουν τουλάχιστον ένα τμήμα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, που είναι κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε, γιατί εμείς θέλουμε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται μόνο για επιπλέον προγράμματα. Λοιπόν, κάποιες από αυτές τις απαντήσεις δεν τις έχω πάρει. Και το τελευταίο που αναφέρατε, για το ελάχιστο ποσοστό για τους διάφορους τομείς και κάποια κράτη-μέλη είπατε ότι δεν το πήραν αυτό πολύ σοβαρά. Έχουν όμως, ε, το έχουν αιτιολογήσει, για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Μπορούμε να τους ε, αποδεχθούμε αυτούς τους λόγους. Νομίζω ίσως και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, κοιτάξτε, στην επιστολή μου, δεν ξέρω αν ήμουν πολύ σαφής, θα ήθελα τώρα να ακουστεί για τα πρακτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ταμεία για τη συμπλήρωση ή για την ενίσχυση των κρατών μελών ε, στην περίπτωση περικοπών στους δικούς τους προπολογισμούς. Ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο έχουν τώρα παρουσιάσει το κάθε πρόγραμμα θα έπρεπε να μας επιτρέπει να δούμε κατά πόσο συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε να έχουμε ένα επίπεδο λεπτομέρειας πιο ενισχυμένο για κάθε κράτος μέλος, ώστε να μπορούμε όλοι μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η Σιλβί Γκυγιόμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη κιόλα γιατί καθυστέρησα να προσπαθήσω κι εγώ να συνεχίσω αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος προηγουμένως. Από ό,τι κατάλαβα ζητήσαμε κάποια διευκρινιστικά στοιχεία και μας ε, δώσατε κάποια παραδείγματα, τρία. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση για ε, τα θέματα αυτά, όπως ε, συγκεκριμένα για το Ταμείο Ενσωμάτωσης και Ασύλου, είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και επομένως είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Όσον αφορά τώρα τα διευκρινιστικά ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε ε, τα ε, στοιχεία αυτά επειδή και εμείς ήμασταν πάρα πολύ ακριβείς κατά την επεξεργασία του κειμένου αυτού. Όσον αφορά την κατανομή των ε, κονδυλίων, είπαμε ότι θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ισότητα. Σας ρωτήσαμε λοιπόν αν, γίνεται, αν γίνονται σεβαστά αυτά τα ελάχιστα ποσοστά και αν υπήρξαν ε, εξαιρέσει για τα ελάχιστα ε, ποσοστά, αν ζητήθηκαν οι εξαιρέσει αυτές, μήπω θα μπορούσαμε συγκεκριμένα να ξέρουμε τι ίδιου εξαιρέσει και για ποιο λόγο ζητήθηκαν. Δεύτερη σειρά ε, διευκρινήσεων για το ζήτημα της επανεγκατάστασης συγκεκριμένα ε, το ερώτημα για το Ταμείο Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης ε, συγκεκριμένα, για να μπορούν τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτήν την προσπάθεια επανεγκατάστασης, αυτό μεταφράστηκε στα εθνικά προγράμματα, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η οικονομική ενίσχυση ε, βοήθησε λίγο τα πράγματα να κινηθούν. Εντάξει, δεν λέω καμία φαινομενική εξέλιξη, αλλά πάση περιπτώσει αν υπήρξε κάποια κίνηση. Και κάτι ακόμη για τις ε, εθελοντικές επιστροφές ε, και τις εξαναγκαστικές ε, επιστροφές. Αυτή η βούληση να προωθήσει κανείς τις εθελοντικές επιστροφές αντί για τις εξαναγκασμένες έχει προχωρήσει, έχει καρποφορήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλάβατε τώρα τι επίπεδο λεπτομεριών μας ενδιαφέρει. Ο Τόμας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση ως εισηγητής αλλά και σκιώδης εισηγητής για διάφορα προγράμματα της προηγούμενης ε, προγραμματικής περίοδου. Πολύ συχνά διαπίστωσε ότι επαναλαμβάνονται τα λάθη και ιδιαίτερα. Τι εννοώ. Δεν λαμβάνει υπόψη την πείρα από την εφαρμογή των, ε, των προηγουμένων προγραμμάτων. Και επίσης πολύ συχνά υπάρχει επικάλυψη, δηλαδή διαφορετικά προγράμματα κάνουν την ίδια δουλειά. Και επίσης δεν έχουμε και κριτήρια για να μετρήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν ε, έχετε ήδη ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Μήπως χρειαστεί λοιπόν ε, μετά από πέντε χρόνια να επανέλθουμε εδώ και να επαναλάβουμε τις ίδιες επικρίσεις προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε προβλήματα με πολλά κράτη-μέλη με τον τρόπο με τον οποίο ε, κάνουν αίτηση και αξιοποιούν αυτές τις πιστώσεις. Κάνετε τίποτα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι... Α, παρακαλώ. Ο κύριος Βόιτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα... Είπατε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βουλγαρία οι περισσότερες πιστώσεις δίνονται για την εθελούσια και μη εθελούσια επιστροφή. Δηλαδή, με ποιο τρόπο ε, γίνονται αυτές οι δαπάνες. Τους δίνουμε κάποιες επιδοτήσεις για να επιστρέψουν θελωσίως ή υπάρχουν άλλα προγράμματα. Και για τις μη εθελούσιες επιστροφές, για αυτές τηρείται το ενωσιακό δίκαιο ή υπάρχουν εθνικές ιδιαιτερότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και την Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσει η Επιτροπή για να μας δώσει κάποιες πρώτες απαντήσεις. Ο κύριος Γκάστελα. Ευχαριστώ για τις ε, πολλές ερωτήσεις σας. Κύριε Βόιτ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία εθελούσες και μη εθελούσες επιστροφές. Κοιτάξτε, εδώ όπως ζητούν οι νομοθέτες να αναβάνει την ευθύνη της η Κομισιόν και επιμένει πάρα πολύ ότι πρέπει να υπάρχει σαφής προτίμηση. Απαιτούμε να προωθείται η εθελούσια επιστροφή. Βεβαίως δεν είναι η μόνη δυνατότητα. Αλλά και πάλι να, να αναφέρω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή τα καταφέρνουμε. Δηλαδή καταφέρνουμε να πείσουμε όπως ακριβώς θέλουμε, να πείσουμε τα κράτη-μέλη να προτιμούν την εθελούσια επιστροφή σε σχέση με την μη εθελούσια. Ίσως στο μέλλον να υπάρχουν άλλα προγράμματα όπου οι εθελούσιες να είναι λιγότερες από τις μη εθελούσιες, αλλά για διάφορους λόγους. Επειδή είναι νέα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, που δεν έχουν ακόμη οικοδομήσει τα συστήματα ασύλου και επιστροφής, που έχουν λιγότερες ε, δυνατότητες, λιγότερη τεχνολογία, λιγότερη πείρα. Αλλά γενικά λέμε και συνεχίζουμε και αδιακόπως και ακούραστα θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι πρέπει να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο η εθελούσια επιστροφή. Θέλουμε λοιπόν να την ευνοήσουμε την εθελούσια, όπως είπα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσο λαμβάνουν ενωσιακούς πόρους πρέπει φυσικά να τηρούν τον ενωσιακό νόμο. Και αυτό το κατέστησα σαφές προς το Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω το κατάλαβαν. για την επανακατάσταση όπως είπε η κυρία Γκυγιόμ γιατί το παρέλειψα και είναι πολύ σημαντικό δεν θέλω να φανώ υπεραισιόδοξος ναι βλέπουμε τα αποτελέσματα υπάρχει ήδη βελτίωση ουσιώδης αύξηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα λοιπόν τώρα ακριβώς επειδή υπάρχει το κίνητρο των χρηματοδοτήσεων των ταμείων Ελπίζω λοιπόν να μην διαψευστώ ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υποσχέσεων και δεσμεύσεων ε, πάμε πολύ καλά μετά να δούμε βέβαια και πώς θα πάει η εφαρμογή. Με συγχωρείτε, ο κύριος Τάμας για το πώς ε, ποσοτικοποιούμε τα αποτελέσματα, πόσο είναι μετρήσιμα, και αν τα κριτήρια μετρησιμότητας. Έχουμε αυτούς τους κοινού δείκτες που είναι κάτι καινούριο και συνεργαστήκαμε πολύ για να έχουμε αυτό τον δίκτυ, το κατάλογο κοινών δικτών για όλα τα κράτη-μέλη για να μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Επιπλέον, επιμείναμε στο μέτρο του δυνατού να έχουμε στοχευμένα αποτελέσματα για συγκεκριμένους δείκτες που θεωρούσαμε ότι είναι οι πιο χρήσιμοι για ορισμένα κράτη-μέλη. Νομίζω θα αυξηθεί λοιπόν η μετρησιμότητα. Λοιπόν, Είπατε επίσης ότι υπάρχει επικάλυψη, ότι χρησιμοποιούνται οι ενωσιακοί πόροι για να καλύψουμε τα δημοσιονομικά κενά των κρατών μελών. Φυσικά το προσέχουμε αυτό, υπάρχει μεγάλος πειρασμός, είναι σαφής, υπάρχουν παντού περικοπές των προπολογισμών, άρα τα κράτη-μέλη μπορεί να υποκύψουν σε αυτό τον πειρασμό. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε άκαμπτοι σε αυτό. Αν κάποια προγράμματα χρηματοδοτούνται ήδη από εθνικού πόρους εν μέρη, τότε να το δούμε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι μας, δηλαδή να χρησιμοποιούνται σκοπίμως για τους στόχους των ταμείων, δηλαδή σε προγράμματα ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, να υπάρχει προσθετικότητα και όχι αντικατάσταση και να μην γίνεται διπλή δουλειά. Αλλά τι θέλω να πω για αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά είναι ετή, έτσι δεν είναι. Αναφερθήκανε συγκεκριμένα προγράμματα. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένα σχέδια. Θα χρηματοδοτήσουμε κατηγορίες προγραμμάτων. Δεν θα ε, λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα σχέδια. Αποφασίσαμε να υπάρχει πιο ευέλικτος προγραμματισμός για να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία, τη σπατάλη. Τη γραφειοκρατία και τη σπατάλη. Είναι πιο ευέλικτα λοιπόν. Κάνουμε πολλές προσπάθειες για να καθορίζουν με το σαφέστερο δυνατό τρόπο τις ενέργειές του τα κράτη-μέλη, αναφερόμαστε μόνο σε παραδείγματα δράσεων, κατηγορίες δράσεων, όχι συγκεκριμένα προγράμματα μια άλλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Δεν θα περιμένουμε πέντε χρόνια για να ασκήσουμε ελέγχου. Κυρία Σίπελ, είναι σημαντικό αυτό. Κάθε χρόνο θα του ελέγχουμε. Και όταν υποβάλλουν ε, του λογαριασμού του. Όταν υποβάλλουν τα προγράμματα θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι έχουν εφαρμόσει προγράμματα. Βέβαια αυτό δεν είναι αντίθετο με αυτό που ζητήθηκε από την πλευρά σα. Πιο συγκεκριμένη δηλαδή πληροφόρηση για το ποιε κατηγορίε δράσεων χρηματοδοτούμε. Βεβαίως θα το κάνουμε. Αλλά να καταλάβουμε όλοι σαφώς ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα με κατηγορίες προγραμμάτων, όχι συγκεκριμένα σχέδια. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αναφέρατε πολύ συγκεκριμένα και σοβαρά θέματα, κυρία Ζήπελ. Λαμβάνουν υπόψη τα ελάχιστα ποσοστά. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Τα λαμβάνουν υπόψη πολύ πιο σοβαρά. Πολύ πιο σοβαρά από ό,τι περίμενα. Πολύ σοβαρά και δεν το είπα στην αρχική μου παρουσίαση. Πάντα μας παρέχουν συγκεκριμένους λόγους για τις εξαιρέσεις και βάσιμους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα τους δεχόμεθα, όχι βέβαια, αλλά μας δίνουν πολύ βάσιμη και συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Ορισμένες φορές τη δεχόμεθα και εδώ είναι και σημαντικό και για εσάς το θέμα. Για αυτό το θέμα θα σας ενημερώνουμε όσο πληρέστερα γίνεται στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή. Όλα λοιπόν τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτά που τους λέμε και κάνουν πολύ και σκληρή δουλειά για να μας εξηγήσουν τι κάνουν. Και μέχρι στιγμής έχουμε πολύ λίγες εξαιρέσεις. Και όπως σας είπα, τις δεχόμεθα αυτές τις αιτήσεις εξαιρέσεων μόνο αν είναι πολύ βάσιμη και μας βρίσκει σύμφωνους, σύμφωνους ή αιτιολόγηση. Μα αυτά νομίζω. Νομίζω ότι απάντησα στι περισσότερε και αν ξέχασα τίποτα, παρακαλώ, υπενθυμίστε μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, δομέ λογοδοσία. Εντάξει, το δεχόμεθα αυτό. Αλλά τα παραδείγματα που έδωσαν οι συνάδελφοι όπω και η κυρία Γκυλιόμ είναι ότι θέλουμε συγκεκριμένη ανάλυση και μάλιστα πληροφορίες ανά κράτος μέλος. Θα θέλαμε λοιπόν μέχρι τον Ιανουάριο, θα το πω στην ε, επιστολή μου, τα μέλη θέλουν ένα επιπλέον επίπεδο λογοδοσίας, γιατί χρειάζεται ένα επιπλέον επίπεδο διαφάνειας για τα προγράμματα αυτά. Και σε αυτή τη φάση δεν έχουμε. Είναι με πολύ χοντρές πινελιές παρουσίασή σας. Δεν επαρκεί αυτό για προγράμματα τέτοιου τύπου. Γι' αυτό θα σας ξαναστείλω την επιστολή μου για να ζητήσω πιο ενδελεχή ανάλυση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσίαση σας σήμερα. Παρακαλώ, κυρία Ζίπελ, μια σύντομη ερώτηση. Μήπως υπάρχει παρανόηση, δεν ξέρω, μήπως είναι γλωσσικό το θέμα. Είπατε ότι κάποιες χώρες ζητούν εξαιρέσεις να μην τηρήσουν αυτά τα ελάχιστα ποσοστά. Είπατε ότι θα πάρετε την περαιτέρω πληροφόρηση στο μέτρο του δυνατού. Μήπως σημαίνει ότι δεν θα τη λάβουμε. Μήπως δεν σας κατάλαβα. Όχι, όχι, είναι γλωσσικό το θέμα. Ήδη σήμερα σας ε, στείλαμε κάποια πληροφόρηση και με συγχωρείτε που δεν το ανέφερα αυτό το σημείο στην ε, εισαγωγική μου παρουσίαση. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όπως σας είπα με βάση την επιστολή του είχα καταλάβει ότι πρέπει να σας δώσω αυτό το επίπεδο προφόρηση αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε το περαιτέρω θα σας δώσω λοιπόν πιο αναλυτική προφόρηση γι' αυτό. Δηλαδή στο μέτρο του δυνατού σημαίνει στο μέτρο του δυνατού βεβαίως. Αλλά να δούμε και σε τι φάση βρισκόμαστε. Ο οριζόντιος κανονισμός καθόρισε ότι θα σας πληροφορήσουμε αναλυτικά και πλήρως στη φάση προγραμματισμού. Αλλά τα προγράμματα ε, υλοποιούνται με βάση τη διαδικασία που σας περιέγραψα. Νομίζω ότι η έκφραση στο μέτρο του Νατού είναι κλασική διατύπωση ε, ενός δημοσίου υπαλλήλου για να ε, προστατευτεί κάπως. Αν εμείς, εγώ, εγώ αρχίσω να τα χρησιμοποιώ, τότε θα πρέπει να φοβηθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε πιο αναλυτική προφόρηση. Θα σας γράψουμε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όλοι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται είναι παρόντες. Ναι, είναι εδώ, τους βλέπω, κάθονται. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να σας τους παρουσιάσουμε. Έρχονται λοιπόν. Έρχονται λοιπόν. Θα σας τους παρουσιάσω. Το επόμενο θέμα είναι μελέτη του Κοινοβουλίου για την Επιτροπή μας νέες προσεγγίσεις και εναλλακτικέ δυνατότητες για τα άτομα που ε, επιδιώκουν διεθνή προστασία. Και εδώ έχουμε τους ομιλητές, θα τους παρουσιάσω. Είναι η Βιολέτα Μορένο Λάξ, που είναι καθηγήτρια λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι συντονίστρια στο, ε, στην πρωτοβουλία για το κέντρο για τους πρόσφυγες του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου και επίσης έχουμε την Κάθριν Κοστέλο που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Andrew W. Μέλλον. Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι γίνονται όλο και μακρύτεροι. Ξέρω γιατί είναι τόσο μακροσκελής. Γιατί όλοι αυτοί που πληρώνουν για τις έδρες έχουν ε, μεγάλα αμερικανικά ονόματα. Είστε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άντρου W. Μέλλορ για διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό δίκαιο στο Κέντρο για Σπουδές για τους Πρόσφυγες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επίσης ε, είστε και διδακτό προσωπικό στο Κολέγιο του Αγίου Αντωνίου. Και έχουμε και μια παρουσίαση από τον κύριο Μίνο Μουζουράκη, ο οποίο είναι στην ε, μονάδα για τις ε, μελέτες για την ε, μη εθελούσια μετανάστευση του Πανεπιστημίου του, της Οξφόρδης, του Κέντρου για τις Σπουδές Προσφύγων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Αυτή η μελέτη ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής μας και το αντίστοιχο τμήμα πολιτικής έδωσε συνέχεια και έχουμε εδώ λοιπόν τους διακεκριμένους ομιλητές μας οι οποίοι είναι οι συντάκτες αυτής της μελέτης θα τους δώσω τώρα το λόγο. Δεν έχουμε κάνει συζήτηση για το άσυλο εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο. Η καθηγήτρια κυρία Κοστέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότομη Μαέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σα για να παρουσιάσω μία μελέτη που έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Δεν χρειάζεται να σα πω πόσο σημαντικέ είναι οι στιγμέ που διανύουμε σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει τη Ευρώπη για του μετανάστε. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία κρίση άνευ προηγουμένου στην Ευρώπη και η κρίση στη Συρία έχει σαν αποτέλεσμα πολλούς εκτομισμένους που κινούνται βασικά σε αυτή την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο γράφτηκε αυτή η έκθεση, δεν γράφτηκε, δεν συντάχθηκε μόνο από εμάς τους τρεις. Θα δείτε ότι υπάρχουν κι άλλοι δύο συντάκτες που δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ. Και υπάρχει και ένα συμβούλιο που, το, και τα ονόματα μπορείτε να δείτε εδώ. Το θέμα δεν είναι τα τρόποι πρόσβασης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λάβατε μια πολύ σημαντική έκθεση από έναν άλλον μελετητή που εξέτασε τις νομικές ε, υποχρεώσεις που έχουμε σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική χορήγηση θεωρήσεων. Θα σας έλεγα το διαβάσετε. Και έγιναν και άλλες μελέτες που εξέτασαν άλλους τρόπους πρόσβαση, διπλωματικό άσυλο, επανα, εγκατάσταση ε, προσφύγων, πρόσφυγες στον καιρό της κρίσης, της δημιουργία μεγαλύτερης εραστικότητας στο καθεστώς που αφορά τις ε, θεωρήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει μια παρουσίαση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας σήμερα το απόγευμα θα γίνει αναφορά στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης από πλευράς της Αυστρίας. Το θέμα της ε, ασφαλούς πρόσβασης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα το δείξουμε όμω αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι το σημείο που θα θέλαμε να το τονίσουμε εισαγωγικά είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν υπάρχει ασφαλή πρόσβαση, το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει παρέκκληση από τη βασική υποχρέωση, την προστασία δηλαδή των ετούντων άσυλο. Με άλλα λόγια, ακόμα και όταν υπάρχει ένα κατάλληλο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ακόμα και όταν υπάρχει ελαστικότητα έτσι ώστε ορισμένοι πρόσφυγες μπορούν να νόμιμα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουν προστασία, οι μηχανισμοί αυτοί δεν αποτελούν υποκατάστατο για την εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων που θα πρέπει να είναι διαρθρωμένες με τον κατάλληλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα αναζήτησης προστασίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι η βάση της ε, ε, εκθεσής μας. Με βάση αυτό κάνουμε ορισμένες υποθέσεις που αφορούν την ε, φύση της αυτόματης, αυθόρμητης αναζήτησης ασύλου. Αυτό οφείλεται στον, στις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που οδήγησαν σε άτακτες, άτακτη είσοδο μεταναστών. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε σε αυτή τη διαδικασία ασύλου. Η μελέτη λοιπόν εξετάζει την προστασία και την υποδοχή. Την πρώτη φάση, αυτά είναι φαινόμενα που συνδέονται μεταξύ τους. Το πώς ε, δηλαδή αναγνωρίζονται οι ε, ε, πρόσφυγες, πώς αυτοπροσδιορίζονται, Όλα αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους αν θέλουμε ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα δύο αυτά σημεία. Μα ζητήθηκε να εξετάσουμε το θέμα της ε, κοινή ευθύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό μιλάει για την επεξεργασία των αιτήσεων, των αιτήσεων ασύλου, αλλά και κοινή ευθύνη σε ό,τι αφορά την αναγνώριση αυτού του καθεστώτος αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζεται αυτό αυτόματα από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα η οποία επεξεργάζεται την αίτηση ασύλου έχει μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστε, ε, τον οποίο το καθεστώ έχει αναγνωριστεί, αλλά δεν μπορούν να συναντήσουν τι οικογένειέ του. Θα θέλαμε πριν να συζητήσουμε νέου μηχανισμού, πριν να μιλήσουμε για κοινή επεξεργασία, πριν να μιλήσουμε για εναλλακτικέ λύσει προ το Δουβλίνο, να εξετάσουμε ποια είναι τα ε, τωρινά προβλήματα. Και πολλά από τα τρέχοντα προβλήματα στο σύστημα σύλλου στην Ευρώπη είναι προβλήματα που έχουμε δημιουργήσει εμεί οι ίδιοι. Οφείλονται στην υπερβολική χρήση καταναγκασμού στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών και των συστημάτων που οδηγεί σε καταστάσεις στις οποίες οι αιτούντες άσυλο δεν την αναγνώριση σε ό,τι αφορά την προστασία τους και ε, και πάρα, πάρα πολλές χώρες πάρα πολύ συχνά δεν τον αγνωρίζουν αυτό, δεν, δεν, είναι, ε, δεν είναι εγγεγραμμένοι, ε, υπάρχουν εκτεταμένες διαδικασίες και πάρα πολύ συχνά χρειάζεται να, μείνουν, να γίνουν ε, Όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε ένα σωστό σύστημα, σε σωστά διαδρομένο σύστημα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επανέλθουμε, να ξεκινήσουμε από τη βάση. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία εξετάζαμε εκτέσεις από διάφορες πηγές. Αυτή η έκθεση ανατέθηκε τον Ιούλιο, την υποβάλαμε τον Σεπτέμβριο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βασιστούμε στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τώρα τα πράγματα ε, και να υποβάλουμε προτάσεις πραγματικά προσπαθήσαμε να, να τονίσουμε το θέμα της υποδοχής στα σύνορα των διαδικασιών και την αναγνώριση συγκεκριμένων αιτήσεων άμεσα. Επίσης συμπληρώσαμε την έρευνά μας με ορισμένες ε, άλλες παράλληλες έρευνες, αυτά θα μας τα εξηγήσει ο Μήνος, ε, μας πίεζε όμως πάρα πολύ ο χρόνος και είχαμε πάρα πολύ λίγες ε, απαντήσεις. Προσπαθήσαμε όμως να πάρουμε το πολιτικό σφιγμό και να καταλάβουμε αν θα ήταν βιώσιμες πολιτικά αυτές οι προτάσεις. Η ουσία λοιπόν της έκθεσης είναι η εξής. Έχει κυκλοφορήσει και μετά ε, έχει ήδη κυκλοφορήσει και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις σας. Στο πρώτο κεφάλαιο Υπάρχουν ορισμένες βασικές πληροφορίες ό,τι αφορά του ίδιου του ετούντε άσυλο και ιδιαίτερα τα όσα περιέχονται στο κεφάλαιο 2. Δηλαδή κάνουμε μία ανασκόπηση του άχθου που αφορά του ετούντε άσυλο στην Ευρώπη. Πριν να δώσω το λόγο στον βουλευτή που θα μιλήσει για τα στατιστικά δεδομένα, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και όταν συζητάμε, θεωρούμε ότι είναι ένα βάρος ε, αυτό είναι μία μάλλον ε, ένας αρνητικός τρόπος να τα βλέπουμε τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι όλη η διαδικασία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τον αριθμό των αιτήσεων αλλά από την ίδια τη φύση των διαδικασιών. Και τονίζουμε ότι σε ορισμένε εκθέσει ε, που συντάχθηκαν στο παρελθόν, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα σε κάθε διαδικασία είναι ο βαθμός στον οποίο είναι καταναγκαστικό αυτό. Αν, ε, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με κράτηση, θα είναι πάρα πολύ ακριβό, αν είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, εάν δεν εφαρμοστεί καλά, τότε δημιουργούνται πάρα πολύ πολύπλοκες διαδικασίες, έφεσης, καταλήγουμε στα δικαστήρια και αυτό αυξάνει το κόστος. Θα θέλαμε λοιπόν να, να προσθέσουμε αυτό το απλό σημείο που αφορά τις κοινέ ευθύνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φαίνεται ότι διερευνούμε τις αναλλακτικές λύσεις στο Δουβλίνο, αλλά πριν να μιλήσουμε για ένα καταμερισμό του, του βάρους, είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε τι βαθμό αυτό το βάρος το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Η Βιολέτα λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέποντας λοιπόν τις στατιστικές, ε, τέσσερα βασικά έτη του κοινού συστήματος ασύλου, 1999, 2004, 2010 και 2014. 2004 ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του κοινού συστήματος ασύλου. Το 2009 είναι το έτος της ε, έναρξης ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας και η ημερομηνία κατά την οποία η Χάρτα Θημελιωδών Δικαιωμάτων κατέστη δεσμευτική. Το 2014 είναι τώρα, μετά την ολοκλήρωση του, της δεύτερης φάσης ε, του ε, κοινού ε, συστήματος ασύλου. Αυτές είναι οι βασικές ημερομηνίες στις οποίες βασιστήκαμε όταν αξιοποιήσαμε τις στατιστικές αυτές. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διακύμανση, αν δει για παράδειγμα κανείς τις τέσσερις στήλε, είναι χαμηλός ο αριθμός, ε, δεδομένου ότι υπήρχαν, ε, υπήρχε και μεγάλη διεύρυνση από 15 ε, σε 27 κράτη-μέλη, είναι αρκετά σταθερός ο αριθμός των μεταναστών και μάλιστα μείωση των αιτήσεων ασύλου παρά το γεγονός ότι αύξηση από, υπήρξε διεύρυνση από 15 σε 28 χώρες, σε γενικές γραμμές ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου παρέμεινε σταθερός. Στατιστικές και πάλι, τα δεδομένα, βλέπετε εδώ τη γραφική παράσταση, στο σύστημα ε, του Δουβλίνου, επειδή υπήρξε καλύτερη κατανομή ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών, βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια ε, διάσταση ε, σε σχέση με το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως η καθηγήτρια Κοστέλο. Βλέποντας λοιπόν τη γραφική παράσταση και πάλι, βλέπουμε ότι έχει παραμείνει ο αριθμός των αιτήσεων ε, ε, αρκετά σταθερός και επειδή έγιναν μεταρρυθμίσεις, επειδή υπήρξε δουβλίνο, αλλαγή από το Δουβλίνο 1 στο Δουβλίνο 2 και μετά από το Δουβλίνο 2 στο Δουβλίνο 3, υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Ε, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, η ε, μεταφορές του Δουβλίνου ε, έχουν, έχουν ε, μειωθεί Υπάρχει μια, ένα μεγάλο κενό μεταξύ των ε, μεταφορών που ζητήθηκαν και των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόστος, τον οποίο να μπορούμε να απομονώσουμε, γιατί υπήρξαν διάφορες δικαστικές προκλήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη υπήρξαν ε, κάποιες πρακτικές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν κάποιες νομικές, ε, κάποιους νομικούς κανόνες, υπήρξε ένα μεγάλο κενό μεταξύ του 12% ε, και των πραγματικών μεταφορών που ήταν περίπου 3% τελικά. Οι μεταφορές δηλαδή που όντως πραγματοποιήθηκαν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καλύψουμε κάποιες από τις ε, ε, αδυναμίες του καθεστώτος του Δουβλίνου και στο κεφάλαιο 3... Αυτό το κεφάλαιο χαρτογραφεί τις βασικές πρωτοβουλίες που αφορούν ε, και τις μεθόδους κατανομής αλλά και τους μηχανισμούς επεξεργασίας για την πρώτη υποδοχή. Όσον αφορά τώρα τις ε, πρωτοβουλίες, ε, τις κοινέ πρωτοβουλίες επεξεργασίας, υπήρχαν προτάσεις ε, οι οποίες έχουν υποβληθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. μέχρι την πλήρη εφαρμογή του μηχανισμού αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρακτικές, ε, κάποια πιλωτικά προγράμματα ΕΑΖΟ για τα διάφορα ε, στάδια της διαδικασίας ασύλου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για ε, περισσότερες κοινέ δραστηριότητες στο μέλλον. Έχουμε επίσης και κάποιες, κάποια εμπειρία από το παρελθόν. Υπάρχει επιτυχής εμπειρία συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάτι το οποίο αν είχε χρησιμοποιηθεί θα είχε ενισχύσει ε, τις ε, δυνατότητές μας ε, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της Mare Nostrum επιχείρησης στη Μεσόγειο. Τώρα, ε, όσον αφορά τώρα τις μεθόδους ε, κατανομής, ε, υπάρχουν δύο τάσεις τις οποίες διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν. Ένα σύστημα κλίδας κατανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο πρότειναν κάποια κράτη-μέλη, αλλά και κάποια ακαδημαϊκοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάλογα με τα μέσα, τις δυνατότητες, με την υποστήριξη βέβαια της αρχής της αλληλεγγύης, συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, προτάσεις ε, αμοιβαίας αναγνώρισης ε, που θα βασίζονται στις υποχρεώσεις της συνθήκης, το άρθρο 78 συγκεκριμένα, για ένα ενιαίο καθεστώς που θα ισχύσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όποιο τρόπο και αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, είτε μια κοινή ε, επεξεργασία ε, είτε ένα σύστημα κατανομής, ένα μηχανισμό κατανομής αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε μία από τις δύο επιλογές, πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο των ετούντων άσυλο, ε, όπως επίσης ε, και ε, τον τρόπο αίτησης και υπηρεσίας. Όσον αφορά το κεφάλαιο 4 για τις νομικούς, τους νομικούς περιορισμούς ε, που είναι δεσμευτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των ε, αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά τις διαδικασίες ε, και το νορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και τις συνθήκες πρώτης υποδοχής. Σε σχέση με την ε, επεξεργασία του ασύλου υπάρχουν κάποιες ε, βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν, ε, όταν ορίζεται, καθορίζεται το καθεστώς του ασύλου. Υπάρχουν τα άρθρα 41 και 47 ε, ή ε, αποφάσεις ασύλου, όχι οριστικές αποφάσεις ε, για το καθεστώς του ετούντος, αλλά για την αναγνώριση, την παραπομπή, την υποδοχή, ειδικέ ανάγκες που μπορεί να έχει ο ετών, αποφάσεις κατανομής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με συνέντευξη ή, εν πάση περιπτώσει, με τον καθορισμό του καθεστώτος του ετούντος άσυλο. βέβαια, υπό τον ε, υπό τον, ε, υπό τον όρο του να υπάρχει πάντοτε δικαιοσύνη και σωστή μεταχείριση κλπ. Ε, το θέμα τώρα της αποτελεσματικής προστασίας που αναφέραμε και προηγουμένως είναι κάτι το οποίο το εξετάσαμε πάρα πολύ. Υπάρχει και νομολογία για το θέμα αυτό. Οι πρώτε λεπτομερεί προδιαγραφέ έχουν να κάνουν με το θέμα του καθεστώτο, κάτι το οποίο πρέπει να μην παρακολύεται ούτε νομικά αλλά ούτε στην πράξη. Επίση, θα έπρεπε να διευκολύνεται η διαδικασία αυτή μέσω ε, αρμόδιο προσωπικού που είναι σωστά κατηρτισμένο για να μπορεί να καθορίσει το καθεστώς, να υπάρχουν ε, υπηρεσίες μετάφρασης και νομική ε, συνδρομή όποτε χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μετά την, μετά την υποβολή αίτησης ε, υπάρχουν, έχουν θεμελιώδη δικαιώματα οι τούντες άσυλο που, που αναγνωρίζονται στη χάρτα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπάρχει και νομολογία του δικαστηρίου. Τρία από, τρία από τα βασικά δικαιώματα αναφέρονται είναι το δικαίωμα στην ελευθερία, στην οικογενειακή επανένωση και στη μία επαναπροώθηση. Ε, η κράτηση ε, μεταξύ των... Βέβαια, η, η, όπως επίσης και η ε, εξαναγκαστική επιστροφή πρέπει να αποτελούν έσχατες λύσεις Τώρα, βάσει της νομολογίας, ε, στην περίπτωση σημάδες ασύρι, υπόθεση σημάδες ασύρι, Η διαδικασία αρχίζει από τη στιγμή της αίτησης, από τη στιγμή δηλαδή της υποβολής αίτησης, ο ενδιαφερόμενος ε, θεωρείται ε, ότι πρέπει να ε, την χάνει μεταχείρισης βάσει της αναθεωρημένης ε, σύμβασης. Νομίζω ότι τις επόμενες διαφάνειες μπορούμε να τις περάσουμε. Βλέπετε στις διαφάνειες πώς πρέπει να γίνονται ε, στο πρώτο βαθμό η εξέταση, η εξέταση των αιτήσεων ε, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση του κάθε ετούντος. Οι αρνητικές αποφάσεις ε, πρέπει να οδηγούν σε διαδικασίες προσφυγής οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα ανασταλτικό αυτομάτως. Πάμε τώρα στην ανάλυση του συστήματος του Δουβλίνου σήμερα. Θα δώσω πάλι το λόγο στον, στην κυρία Κοστέλο. Αλλά αυτό που εμείς διαπιστώσαμε με τη μελέτη μας, αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το σύστημα και είδαμε το ανθρώπινο κόστος του συστήματος του Δουβλίνου αλλά και το οικονομικό κόστος και το νομικό κόστος. Όσον αφορά το ανθρώπινο κόστος, ε, φάνηκε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που ε, ε, επιδεινώνονται από αυτούς που, που, που δείχνουν ότι ε, φάνηκε ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί που καλύπτονται από το σύστημα του Δουβλίνου και τελικά ε, υφίστανται τραύματα στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής Δεν υπάρχουν όμως επαρκή στοιχεία αυτή τη στιγμή για να γνωρίζουμε λίγο ε, περισσότερα. Πριν ε, δώσω και πάλι το λόγο στη ε, συνάδελφο, αυτό που θα ήθελα να πω για την αξιολόγηση του συστήματος είναι το νομικό κόστος, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει επαρκής εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας, κάτι το οποίο σήμαινε νομικές προκλήσεις σε, διάφορο, σε διάφορα επίπεδα. Ε, έχει φτάσει στα ανώτερα δικαστήρια ε, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και αφορούσε ακριβώς την μη εφαρμογή των, της τρέχουσας νομοθεσίας. Λόγω ε, μη συμμόρφωσης της μεταφορές υπό το σύστημα του Δουβλίνου με την αρχή της μη επαναπροώθησης και η μελέτη διαπιστώνει ότι έχει φτάσει η στιγμή αναθεώρησης του συστήματος του Δουβλίνου και ενδεχομένως μιας αναθεώρησης του τρέχοντος ε, συστήματος. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το σύστημα του Δουβλίνου και ότι μια σειρά από κράτη-μέλη το εφαρμόζουν ε, ευχαρίστως για διάφορους λόγους. Θέλουμε λοιπόν ε, ένα νέο σύστημα που το αποκαλούμε Δουβλίνο χωρίς καταναγκασμό και επειδή πρέπει να αφήσουμε και χρόνο για ερωτήσεις στην έκθεση αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο με την σημερινή του δομή θα μπορούσε το Δουβλίνο να εφαρμοστεί για να μειωθεί το κόστος για τους ανθρώπους αλλά και το δικαστικό κόστος το οποίο ε, δημιουργεί ε, πολλές αμφισβητήσεις από πλευρά των ετούντων άσυλο. Γιατί μερικές κυβερνήσεις επιμένουν να γίνονται μετακινήσεις ή μεταφορές ε, με βάση το σύστημα του Δουβλίνου παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίε σε μια σειρά από κράτη-μέλη είναι ακατάλληλε. Κάτι άλλο που είπαμε στην έκθεση είναι να περάσουμε από τις νομικές αρχές που ήδη αναφέραμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο, μια σειρά από αρχέ που θα πρέπει να είναι η βάση οποιασδήποτε αλλαγής του συστήματος. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε πολυπλοκότητα ούτε ε, μία αναγκαίος καταναγκασμός. Γι' αυτό θέλαμε να αναφέρουμε τους βασικούς ε, όρους ε, ενός νέου συστήματος κατανομής θα πρέπει να ληφθούν αυτοί οι όροι υπόψη. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ευάλωτοι οι αιτούντε άσυλο και δεν πρέπει να είναι ποινικοποιημένη οποιαδήποτε προσέγγιση των προσφύγων. Αυτό είναι κάτι που το εγγυάται η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και επίση χρειάζεται λογοδοσία, διαφάνεια και έμπειρη γνώμη και πρέπει επίσης να εμπιστεύονται όλοι οι συμμετέχοντες της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Μια πρώτη σοβαρή δυσχέρη είναι ότι η πρώτη επαφή μεταξύ των ετούντων και των αρχών δεν δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό προτείνουμε κάπως ε, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ούτως ώστε η διαδικασία ασύλου να είναι σύντομη, να αναγνωρίζεται σύντομα όποιος έχει βάσιμους λόγους και να μπορέσουν οι πρόσφυγες αυτοί να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους και να ενταχθούν στην κοινωνία. Ο συνάρφος μου ο Μήνος έκανε τις στατιστικές μελέτες και θα σας εξηγήσει μερικά από τα απορίσματα ε, πιο λεπτημερός και μετά θα καταλήξουμε και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ Κάθριν. Καλημέρα σε όλους ε, μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία που απετέλεσαν τη μεθοδολογία μας. Όπως είπε η Κάθριν, λόγω του χρονικού περιορισμού της μελέτης, είχαμε ένα περιορισμό αριθμό απαντήσεων, οπότε είχαμε απλώς μια γενική γεύση των θέσεων και όχι τη δυνατότητα να αντλήσουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Στο βαθμό που μπορούμε να βασιστούμε στις συνεντεύξεις και στην έρευνά μας, βλέπουμε όχι χάσμα αλλά ποικιλία απόψεων σε σχέση με το εφικτό και το πολιτικά επιθυμητό μέτρων όπως εναλλακτικά μέτρα κατανομής ε, ε, και ε, μεταφοράς των ε, ζητούντων άσυλο. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις με ορισμένους οι οποίοι υποστηρίζουν τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και θα οδηγήσουν σε πιο συνεργατική και αποτελεσματική προσέγγιση στο σύστημα ασύλου. Και από την άλλη πλευρά οι δικές μας προσπάθειες μέσα στο 2014 φάνηκαν σαν θετικά παραδείγματα για αυτήν την αντιμετώπιση. Υπήρξε όμως αντίθετη άποψη από ορισμένα που θεώρησαν ότι στην τωρινή ε, κατάσταση του συστήματος ασύλου βρήκανε κάπως πρόορη αυτήν την ε, πρωτοβουλία και ορισμένα νομικά εμπόδια υπάρχουν, όπως παραγωγός η πρόσβαση σε εθνικά συστήματα τράπεζα δεδομένων για τους ε, ετούντος άσυλο και προβλήματα με το γλωσσικό, με γλωσσικά καθεστώτα κτλ. Όπως ανέφερε η Κάθριν προηγουμένως, υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τη διατήρηση του συστήματος του Δουβλίνου ως το σύστημα κατανομής των αιτήσεων για άσυλο αυτή τη στιγμή, αναμένοντας την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου 3 που ενεκρίθη πρόσφατα, ενώ συγχρόνως υπάρχει η άποψη ότι το Δουβλίνο θα πρέπει εν καιρό να αντικατασταθεί με ένα μηχανισμό που θα αποτελεί μια κλίδα κατανομής και θα υπακούει σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των των ασύλου Επίσης είχαμε μια ανάμεικτη αντίδραση στην ιδέα της αμοιβαίας αναγνώσης των θετικών αποφάσεων ασύλου. Από τη μία πλευρά, ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό είναι το επόμενο λογικό βήμα για το σύστημα ασύλου, κάτι το οποίο θα οδηγήσει, θα πρέπει να είναι κομμάτι της δεύτερης φάσης εναρμόνισης. Άλλοι το θεωρούν ότι είναι πρόωρο και θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί το μόλις εγκριθέν και εκτιμένο και να περιμένουν μέχρι ότου τα διαφορετικά συστήματα ασύλου μπορέσουν να φτάσουν σε επίπεδο εναρμόνιση προτού αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ακόμα και το ζήτημα τη της αμοιβαία ε, αναγνώριση τη χάνει διαφορετικών ερμηνεών από τα κράτη-μέλη. ορισμένα κράτη-μέλη, η αμοιβαία αναγνώριση των θετικών αποφάσεων για άσυλο και η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ετούντων ασύλου που την χάνουν ε, προστασίας και επικουρικής προστασίας αυτό δεν θα έχει αυτόματο χαρακτήρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούν οι πρόσφυγες που έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους ελεύθερα σε άλλα κράτη-μέλη για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι στο βαθμό που μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα το πολιτικό οποίο αυτή τη στιγμή είναι κάπως ανάμεικτο και υπάρχουν διαφορετικές και αποκλίνουσες κατευθύνσει. όλα αυτά τα θέματα θα απαιτήσουν πιο προσεκτική και λεπτομεριακή συζήτηση προτού μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Και νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε τα ερωτήματά σας, αν έχετε. Εντάξει. Ναι, εγώ θα αποφασίσω τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι συνάδελφοι. Αλλά υπάρχουν και δύο άλλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, συζητήσουμε διάφορες πλευρές ε, της πολιτικής ε, ασύλου, για παράδειγμα επανεκατάσταση. Και το άλλο είναι η εφαρμογή του υπάρχοντος ε, πακέτου ασύλου. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτήν την έκθεση που υπερβαίνει τις συνήθεις εκθέσεις που μας κάνουν οι υπηρεσίες μελετών του Κοινοβουλίου είναι ότι προτείνεται ένα νέο πρότυπο Δουβλίνο χωρίς εξαναγκασμό. Πολύ ενδιαφέρον. λέτε ε, μάλιστα συγκεκριμένα Δουβλίνο χωρίς ξαναγκασμό και χωρίς ε, Λέτε ότι ορισμένες από τις πολιτικές ε, έχουν και ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς ο εξαναγκασμός. Υπάρχει λοιπόν και αποτροπή και εξαναγκασμός. Το βασικό θέμα όμως για το οποίο θέλουν να θα ήθελα ενδεχομένω να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, είναι ότι αν θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε το Δουβλίνο πρέπει να θέσουμε το βασικό πολιτικό ζήτημα. Δεν θα υπάρξει κατανομή εάν δεν θέσουμε το βασικό ερώτημα προς τα κράτη-μέλη. Θα αλλάξουν τη βασική τους προσέγγιση τα κράτη-μέλη. Γιατί όπως βλέπουμε οι περισσότεροι ετούντες άσυλο καταλήγουν σε τέσσερις χώρες. Ενώ έχουμε 28 κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ουσιώδης πολιτική ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Πολλοί είχαν ζητήσει αυτή η μελέτη, είχαν ζητήσει αυτή τη μελέτη. Οπότε να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Ντεγιόν, ο Ντένις. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου ζήτησε την πολιτική ομάδα. Ωραία λοιπόν που την έχουμε. Σωστά λέει η μελέτη αυτή ότι ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση στα κράτη-μέλη το σύστημα του Δουβλίνου τα έχει φτύσει. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί σε όλο και λιγότερα κράτη-μέλη. Οι μεταφορές ετούν τον άσυλο από, το ένα κράτος μέλος, από ένα κράτος μέλος σε άλλο είναι ελάχιστη και το κόστος και το δικαστικό κόστος και το κόστος ε, για τους ε, ανθρώπους είναι πολύ ψηλό. Γι' αυτό στην ομάδα μου έχουμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση για το μέλλον του συστήματος ασύλου και το στοιχείο του καταναγκασμού είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Τα καταλαβαίνω, τα σέβομαι όλα αυτά. Καλό να κάνουμε τη συζήτηση. Ωστόσο, ωστόσο, όταν ζητήσαμε να γίνει μια μελέτη, όχι μόνο κάναμε μια σύντομη αιτιολόγηση, αλλά προσθέσαμε και ένα σύντομο κείμενο που λέει ότι θα θέλαμε να μάθουμε ιδίω πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των πολύ μακρών συνόρων που έχουμε, που είναι δύσκολο να τα επιτηρούμε και μετά πώς θα μπορέσουμε κοντά στα σύνορα, αλλά εντός της ε, επικράτεια τη Ένωση να έχουμε ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχή προσφύγων, όχι ελληνικά, ιταλικά, ευρωπαϊκά. Με όλε τι εγγυήσει για την υποδοχή, για την εξέταση των αιτήσεων, την πρώτη εξέταση. Και είναι πολύ περίπλοκο να έχουμε τέτοια κέντρα. Γιατί πρέπει να δούμε ποιος θα έχει την ευθύνη, ποιος θα έχει την νομική ευθύνη για τις ε, ε, ε, εφέσεις, για την επιστροφή αυτών των οποίων απορρίπτεται η αίτηση πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πιο περίπλοκες αιτήσει. Τα θέσαμε όλα αυτά στην, ε, στο τμήμα πολιτικής και δεν βλέπω απαντήσεις. Είναι κάπως απογοητευτικό αυτό. Γιατί Έλπιζα ότι θα μπορούσαμε να πούμε κοιτάξτε δεν λειτουργεί το σύστημα, δεν είναι ούτε ανθρωπιστικό ούτε αποτελεσματικό είτε να πούμε ναι είναι μια καλή βάση επί της οποίας ε, μπορούμε να βασιστούμε για να προχωρήσουμε. Αλλά δεν βλέπω τίποτα από αυτά στη μελέτη. Μόνο λίγες ε, σελίδες ασχολούνται από τις 100 σελίδες ε, της μελέτης. Αν είναι λοιπόν η έκθεση. Βεβαίως έχει ενδιαφέροντα χρήσιμα στοιχεία. Ωραίο σύνθημα Δουβλίνο χωρίς καταναγκασμό. Αλλά άμα διαβάσετε τι σημαίνει, σημαίνει τα κράτη-μέλη θα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να μεταφέρουν ε, ετούντε ε, προ άλλα κράτη-μέλη όπου ξέρουν ότι δεν είναι καλές συνθήκες υποδοχής. Αυτό δεν είναι και πολύ σοβαρή αλλαγή, ελάχιστη αλλαγή. Παραμένει στην ουσία το σύστημα Δουβλίνου, ενώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι τόσο τεράστια τα προβλήματα που θα έπρεπε να μας οθήσουν να ξεπεράσουμε το Δουβλίνο και να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα κοινό σύστημα ασύλου και τι επιπτώσεις θα είχε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των ερευνητών. Ναι, πολύ απευθείας ερωτήσεις. Είναι πραγματικά πολύ άμεσες οι ερωτήσεις. Οπότε βεβαίω να απαντήσουμε πρώτα σε αυτές τις πολύ απαιτητικέ ερωτήσεις από όλους τους συναδέλφους και θα σας παρακαλέσω να συνοψίσετε στο τέλο. Σιλβί Γκυλιόμη, επόμενη. Παρακαλώ. Θα πρέπει να πω ότι είμαι κάπως, λίγο, κάπως μπλεγμένη δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς λέτε. Άκουσα τον πρόεδρο που έκανε μια ανακεφαλαίωση λέγοντας ότι είστε υπέρ ενός νέου Δουβλίνου. Ο κύριος Ντεοντιγιόν λέει ότι μιλάμε για ένα βελτιωμένο Δουβλίνο, μια βελτιωμένη έκδοση. Θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Συμφωνώ ότι πριν να μιλήσουμε για εναλλακτικέ λύσεις θα πρέπει να βασιστούμε στα ήδη υπάρχοντα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα θίξατε, η βάση των δυσκολιών σε ό,τι αφορά το κοινό καθεστώς ασύλου είναι το Δουβλίνο, γιατί ξεκινάμε από την αρχή ότι όλα τα συστήματα είναι ίσα, πράγμα που δεν συμβαίνει, ισότιμα. Ζητάμε αυτή τη μεταφορά 12% στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται ένα 3%. Ε, ε, στην ουσία αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να αναγνωρίσω στα συμπεράσματά σας κατά πόσον θα πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε το μηχανισμό αυτό ή αν θα πρέπει να θέσουμε καλύτερα σε εφαρμογή τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Εγώ τουλάχιστον ε, έτσι το κατάλαβα, γιατί κλείθηκα να πω τη γνώμη μου, κατάλαβα ότι υπάρχουν κι άλλα μέσα. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας διαφωτίσετε, θα μπορούσατε να μας πείτε αν θα πρέπει να ανατρέψουμε το σύστημα, να δημιουργήσουμε νέα κριτήρια ή να βελτιστοποιήσουμε το ήδη υπάρχον. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι αυτό σαφώς θα μπορούσε να επηρεάσει το ευρύτερο πεδίο του ε, σε ό,τι αφορά το κοινό καθεστώς ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. <clears throat> Uh, Μικρόφωνο παρακαλούμε have made Δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι οι δύο προλαλήσαντες αναφέρθηκαν σε αυτό που σκέφτηκα και εγώ να πω. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι ακόμα και για μας που γνωρίζουμε αυτή την πολιτική που αφορά το άσυλο, και τον τρόπο που διαρθρώνεται, που σε εφαρμογή μετά τη συνθήκη Λισαβόνα, ακόμα και για μα, είναι πραγματικά δύσκολο. <coughs> Γιατί πραγματικά το όλο θέμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Όταν προσπαθήσαμε στην, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πριν από τις εκλογές του Μαΐου, όταν προσπαθήσαμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι η πολιτική του ασύλου έχει αναθεωρηθεί, έχει ανανεωθεί μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το μήνυμα αυτό δεν έγινε αντιληπτό και δεν έγινε και πιστευτό. Γιατί οι διαφορές οι διαφορετικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από διάφορες χώρες μέλη με εντελώ τερογενείς τρόπους εφαρμογής ε, της πολιτικής ασύλου ήταν η αιτία. Θέλω να καταλάβω με τι τρόπο θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το περιθώριο ελιγμών που έχουν οι χώρες μέλη σε ό,τι αφορά την εθνική εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος ε, για να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα, αυτή την αδυναμία. Υπάρχει η δυνατότητα να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πραγματικά ευρωπαϊκή δύναμη κρούσης η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι το όλο πακέτο νομοθεσία για περί ασύλου θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από τι χώρε μέλη και θα εφαρμοστεί σε ένα συνεπή Με λίγα λόγια, κάτι λιγότερο ετερογενές που να αφήνει πολύ λιγότερο περιθώριο για παρεκκλήσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι αυτό ένα ενδεχόμενο. Θα μπορούσε αυτό να γίνει τα πλαίσια της συνθήκη της Λισαβόνας ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία, μιλάμε για την εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Η Σισίλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ε, μελέτη που μας παρουσιάζεται. Τον Ιούνιο, όταν εγκρίναμε το ε, κοινό σύστημα ασύλου, καταλάβαμε ότι θα ήταν δύσκολη η εφαρμογή του και ε, επίπονη για κάποια Νομίζω όμως ότι θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερων κανόνων και καλύτερων εγγυήσεων ε, για την διαδικασία αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε και να θεωρήσουμε ότι τα καταφέραμε να βρούμε την τέλεια λύση όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μια τέλεια λύση. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα τα επόμενα βήματα προκειμένου να βελτιώσουμε και να βρούμε λύσεις για προβλήματα τα οποία δεν είχαμε προβλέψει τη στιγμή που επεξεργαζόμασταν το πακέτο και η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να προβλέψει 100% πάντοτε. Οπότε ελπίζουμε η μελέτη σας να μας διαφωτίσει, να μας βοηθήσει να βρούμε κάποιες λύσεις. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για τον κανονισμό Δουβλίνο 3 και τώρα είμαι εισηγήτρια για την αλλαγή στο άρθρο 8 του Δουβλίνου, δηλαδή τους ασυνόδευτους ανηλίκους ε, μετά την απόφαση ε, του δικαστηρίου ε, MA και άλλοι την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα δεν είναι ένα εργαλείο αλληλεγγύης, μας δίνει, τα αποτελέσματά του δεν είναι βιώσιμα ούτε για τα κράτη-μέλη. Μόνο λίγες περιπτώσεις ε, ε, Δουβλίνου, όπως ανέφερε και η συνάδελφος ε, Σιλβί ε, έχουν ολοκληρωθεί. 3% είπαμε μεταφορές υπήρξαν στο πλαίσιο του Δουβλίνου. Είπατε όχι εξαναγκασμός. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τις διακριτικές ρήτρε για να υπάρχει καλύτερη κατανομή ευθύνη, όπως επίσης και να λαμβάνονται υπόψη προτιμήσεις των ετούντων άσυλο. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία απολύτως ένδειξη ότι τα κρατη θα κάνουν κάτι τέτοιο στην πράξη. Τουναντίον, έχουμε δει ότι οι ρήτρε διακριτική ευχέρεια ε, χρησιμοποιούνται σπανίω ή και καθόλου. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα το κάνουν αυτό εθελοντικά με τη θέλησή του. Ακόμη και στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, μπορούμε να δούμε καθαρά ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν τη δυνατότητα μεταφορών ακόμη και των ανηλίκων, ως το δυνατόν πιο ανοιχτή. Πώς μπορούμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι μια βιώσιμη λύση για το μέλλον, ότι χρειάζεται αλλαγή και ότι η αλλαγή αυτή είναι είναι απαραίτητη, είναι επίγουσα. Ε, τα κράτη-μέλη, ε, πώς μπορούμε να μην υπάρχει εξαναγκασμός όταν έξι κράτη-μέλη σήμερα ε, μεταχειρίζονται πάνω από 60% όλων των αιτήσεων ασύλου ολόκληρης της Ένωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε βελτιώσουμε την κατάσταση. Ίσως κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα το ε, οποίο ε, θα είναι ε, υπό τη διαχείριση του ΕΑΣ, όπως και ο συνάδελφος De Jong μας είπε, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα αυτό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να δούμε αυτή τη λύση ως πιθανή. Σεσίλια, όσο μιλούσες, ρωτούσα ποιε είναι οι δυνατότητες συνέχισης, αλλά είμαι βέβαιη ότι η δουλειά συνεχίζεται από τους ε, συντάκτες της ε, μελέτης. Ε, θα συνεχίσει η δουλειά τους, παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνά τους. Απλώς, για να απαντήσω σε αυτό που είπες, το είπα αυτό. Ο Τζόζεφ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη και πολλά καθησυχαστικά στοιχεία περιέχει. Θετικό είναι ότι είναι δυνατόν το σύστημα αυτό να έχει μη αποτρεπτικό, μη καταναγκαστικό χαρακτήρα. Όμως νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα είναι κάτι που δεν ήταν αντικείμενο της μελέτης σας. Δηλαδή το θέμα, το ερώτημα, ποια είναι τα σημεία εισόδου στο σύστημα γιατί χωρίς μια μεταρρύθμιση αυτών των σημείων πρόσβασης εκεί που γίνεται η πρώτη εξέταση αν γίνεται με αρκετά ανθρωπιστικούς λόγους δεν ξέρω πώς θα το αποκαλέσουμε αυτό, το σημείο υποδοχής, είναι βασικό. Δηλαδή το σημείο εισόδου, εάν και κατά πόσο στα σημεία εισόδου υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το δούμε γενικά στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής, διότι βεβαίως αν έχω τη δυνατότητα, αν δεν έχω τη δυνατότητα να εισέλθω νομίμως σε μια χώρα, τότε βεβαίως ε, παραφορτώνουμε το σύστημα ασύλου. Βεβαίως ε, αποκαλέσατε αυτή την πολιτική, πολιτική που βασίζεται στα στοιχεία. Είναι λοιπόν πολύ θετική η πρότασή σας, αλλά νομίζω ότι δεν θα μας αρκέσουν αυτές οι πολιτικές που να βασίζονται στα στοιχεία. Δεν θα μας αρκέσουν για να λύσουμε το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε πολιτική λύση και το σώμα μας πρέπει να σκεφτεί τι ακριβώς θέλουμε να αντικαταστήσει το Δουβλίνο. Διότι τώρα ε, το Δουβλίνο είναι η μόνη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παλεύουμε ε, να βγούμε, αλλά μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε μια σαφή πολιτική λύση. Και αυτό είναι το δικό μας καθήκον ως εκπροσώπων του λαού, να διατυπώσουμε τις προϋποθέσεις για αυτή την πολιτική λύση. Πρόεδρος. Αυτοί ήσαν οι ομιλητές. Ενδιαφέρον είναι αυτό που υπόθηκε ότι χρειάζεται πολιτική λύση παρά αυτά που είπε ο Ντένις Τεγιόγκ όπου είπε ότι είχε ζητήσει ε, κάτι και τελικά η μελέτη τι περιέχει. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να εκπονήσει κανείς μια τέτοια μελέτη όπως είπε και η κυρία Βίξτρομ και η κυρία Γκυγιόμ και άλλοι συνάδελφοι και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον τομέα αυτό, ένα από τα προβλήματα είναι η εφαρμογή. Και πίσω από τα προβλήματα εφαρμογής υπάρχουν πολιτικά θέματα. Είπατε ότι υπάρχει περιπλοκότητα, ότι είναι φραγμός η περιπλοκότητα. Και αυτό πολιτικό θέμα είναι, όπως είπε και ο Γιώζεφ, ο τελευταίος ομιλητή. Τώρα δεν θέλω να εκφράσω ε, κρίση επί της αξίας, ε, αλλά η εφαρμογή και η αποτίμησή της είναι πολύ δύσκολο να περιληφθεί σε μια έκθεση. Ο Ντένις Τεγιόν είπε ότι θελήσαμε να μας πείτε τι εναλλακτικέ λύσεις, συγκεκριμένες ερωτήσεις, πώς μπορούμε ως νομοθέτες να παρακάμψουμε το πρόβλημα. Τι εναλλακτικέ στρατηγικές έχουμε. Γιατί πρόκειται για άτομα, για ανθρώπους που έχουν μπει στο σύστημα τώρα, προσπαθούν να λάβουν άσυλο. Λοιπόν, αυτό να αντιμετωπίσετε πρώτα απ' όλα καθαρά. Τι ζητήθηκε και τι περιέχει η έκθεση. Και για το διαδικαστικό τώρα θέμα. Βεβαίω είναι η τελική σας έκθεση και περιέχει πολύ πολύτιμε πληροφορίες. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε την έκθεση βεβαίως, αλλά στην ε, περαιτέρω εργασία σας θα θέλαμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας γιατί φυσικά θα δώσετε συνέχεια σε ορισμένα από αυτά που ανέφεραν συνάδελφοι και η εφαρμογή είναι ο κρίσιμος τομέας γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με το πακέτο. Τα κράτη-μέλη δεν το εφαρμόζουν όπως προβλέφθηκε. Λοιπόν, ε, μήπως να ξεκινήσετε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μείνει χρόνος και τους συναδέλφους. Ξεκινώντας από αυτό που είπε ο κ. Δεγιόν, όταν εξετάσαμε το θέμα της κοινή διαδικασίας, σε ό,τι αφορά τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ασύλου, είχαμε κατά νου το γεγονός ότι ανεξάρτητα από το πώς θα δημιουργεί το αυτό το κέντρο, θα βρισκόταν για την έδρα του σε μία χώρα μέλος και θα υπόκειτο όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο της χώρας μέλους. Όταν σκεφτήκαμε τη θεσμική διάσταση, κάτι που καταλάβαμε από εμπειρικέ μελέτε είναι ότι η ολιστική προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, πολλές οικονομίες. Η, επίσης, ε, μια πολυκλαδική προσέγγιση, μια προσέγγιση από πολλούς φορείς. Ε, πολύ συχνά σε μικρά κέντρα υποδοχής εμπλέκονται και ΜΚΟ καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εκεί όμως δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία οι αιτούντες άσυλο νιώθουν πολύ πιο άνετα. Υπάρχουν, ε, γίνεται αφορά σε πολλές εμπειρικές εργασίες στη μελέτη Διστάζουμε όμως να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα κέντρα. Εδώ μιλήσαμε για νομική εφαρμοσιμότητα, γιατί εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες. Μιλήσαμε και για πρακτικά θέματα που αφορούν τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής. Αυτά είναι θέματα που προσπαθούμε να επιλύσουμε δημιουργώντας ένα σύστημα που θα μπορούσαν να οι άσυλο είναι ευκολότερο να εμπιστευτούν ένα μικρό κέντρο υποδοχή. Επιτρέψτε μου να πω κάτι γενικό. Είναι μεταβατική η κατάσταση του ετούντο άσυλο. Ενδεχομένω ε, διαρκεί ένα μικρό, σύστημα, ε, ένα μικρό διάστημα μέχρι που να αναγνωριστεί το, ε, ένα συγκεκριμένο καθεστώ που απαιτεί προστασία. Όπως είπαμε, οι αποφάσεις για το άσυλο δεν διευκολύνουν ε, την, κινήση, την μετακινήση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς κινηθήκαμε προς μια κοινή αναγνώριση των αποφάσεων περί ασύλου. Ε, πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα έγγραφο γι' αυτό. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν τις κοινέ διαδικασίες, πιστεύουμε ότι έχει κάποιο νόημα όταν κινηθούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό και για την ώρα δεν γίνεται αυτό. Συνεπώ, το θέμα δεν είναι ότι προσπαθήσαμε να ε, μην υιοθετήσουμε μια καινοτόμο σκέψη. Έχουμε απόλυτη συνείδηση όμω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που λειτουργούν σε μικρή ε, κλίμακα. Η αίτηση ασύλου θα πρέπει να είναι μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία που να δημιουργεί προβλήματα εφαρμογή. Και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετε πολυπλοκότητε. Αν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ενό ευρωπαϊκού και ενό τοπικού κέντρου υποδοχή, θα πρέπει να δούμε ποιε αιτήσει θα διέχεται το αίμα, ποιε το άλλο. Και θα πρέπει να αποφασίσει ένα ολόκληρο γραφειοκρατικό σύστημα. Τα ευρωπαϊκά νομικά μέτρα ε, έχουν ορισμένα αδύνατα σημεία. Θα θέλαμε λοιπόν να, να, να πούμε ότι το θέμα του, του ευάλωτου χαρακτήρα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει επιπλέον ε, ε, περιπλοκές. Όταν εξετάσαμε τα μοντέλα της κοινή επεξεργασίας, μερικά από αυτά φαίνονται τοπικά. Το να υπάρχει δηλαδή μια ενιαία αρχή σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε και η άποψη ότι δεν θα έχουν πρακτικό όφελος πέρα από τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Υπάρχουν ορισμένες πιλωτικές μελέτες για την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων. Το θέμα είναι να δούμε ποιος θα ωφεληθεί. Σε κάθε περίπτωση δεν μας απασχολούσε αυτό σε αυτή την έκθεση. Συνάδελφοί μου θα μπορούσαν να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά Ε, εγώ μιλάω για θέματα γενικά. Υπάρχουν ορισμένα θέματα εφαρμογής και το κενό που υπάρχει στον τομέα τη εφαρμογή. Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορε απαντήσεις που θα μπορούσαμε να δούμε. Τα ε, νομικά μέσα εφαρμογής είναι καινούργια, δεν υπάρχει διαδικασία εφαρμογής. Υπάρχει ένα καινούριο ε, δημοσιονομικό εργαλείο το σύστημα τροφοδοτείται και με άλλους πόρους για να βοηθηθούν τα συστήματα που έχουν πιο αδύναμα συστήματα. Πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο ιδιαίτερα σε επίπεδο υποδοχής το να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών για τον έλεγχο της δαπάνης των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ε, πρόσφατη απόφαση του, ε, ε, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έγινε μια αναφορά στην Ιταλία. Πάρα πολλέ φορέ ο Παναπατρισμό θεωρείται τιμωρία. Υπάρχουν ορισμένα καλά οργανωμένα κέντρα υποδοχής στην ε, Ιταλία και είναι αυτά τα κέντρα στα οποία συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών και εκεί οι αιτούντες άσυλο μπορούν να τύχουν κάποιας, ε, κάποιας βοήθειας και να ε, ενημερωθούν για τις νομικές διαδικασίες. Αυτά φαίνονται κοινότοπα, αλλά είναι τα, τα πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ε, ορισμένα κέντρα μαζικής υποδοχής ε, στην Ευρώπη παρέχουν βοήθεια, αλλά η βοήθεια πρόκειται μόνο από την ε, κυβέρνηση και αφορά ε, τούντες άσυλο και το πώς μπορούσαν να επαναπατριστούν θα μπορούσαμε ε, να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα με αυτές τις μεθόδους και νομίζω ότι αν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των κέντρων υποδοχής, μία προϋπόθεση θα έπρεπε να είναι η πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών. Και βέβαια να υπάρχει συμμετοχή πολλών φορέων. Και αναφερθήκαμε και σε ορισμένα πρακτικά θέματα, το πώς ε, ε, εφαρμόζεται, τι γίνεται στην πρώτη φάση της υποδοχής. Το τελευταίο σημείο, σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικέ λύσεις στο Δουβλίνο, νομίζω ότι υπάρχουν δύο πτυχές εδώ. Το ένα αφορά τα κριτήρια κατανομής και ε, σε αυτό αναφερθήκαμε περιληπτικά. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής, δηλαδή τα διάφορα κριτήρια για να αξιολογήσουμε τον αριθμό των ετούντων άσυλων για κάθε κράτος. Εδώ θα ήθελα να μιλήσω για πολιτικές συμφωνίες, γιατί αν θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πολιτικέ συμφωνίε. Οι εθνικέ κυβερνήσει δεν ελέγχουν μόνε τους αυτό το θέμα. Εδώ μιλάμε για καθεστώ συναπόφαση. Οι εθνικέ κυβερνήσει μπορεί ζηλότυπα να κρατάνε την ε, πολιτική μετανάστευση, αλλά είστε συν ε, Θα θέλαμε επίση να τονίσουμε, ακόμα και αν υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια κατανομή, θα έπρεπε να αποφασίσουμε ποιο πηγαίνει πού. Και τίθεται και το ανθρώπινο ερώτημα. Το ποιος πάει πού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη είναι ότι πάρα πολύ συχνά υπάρχει παράνομη μετανάστευση, ε, υπάρχουν ε, ε, ε, ε αυτοί που αυτο ειναι ιδιαιτερα σημαντικο η πραγματικοτητα σημερα στην ευρωπη ειναι οτι παρα πολυ συχνα υπαρχει παρανομη μεταναστευση ε υπαρχουν αυτοι που συγκαλυπτουν την παράνομη μετανάστευση, υπάρχει παραπληροφόρηση. Αν στην πρώτη υποδοχή υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση, εάν ενημέρωνε η κοινωνία των πολιτών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των αιτήσεων ε, ασύλου, ε, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Είναι σε αυτό το σημείο γιατί υπάρχουν, γίνονται γραφειοκρατικές επιλογές. Ενδεχομένως δίνουμε την εντύπωση ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να υποβάλουμε ρεαλιστικές προτάσεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη για το θέμα των κέντρων ασύλου, των ευρωπαϊκών. Νομίζω ότι γι' αυτό το αφήσαμε εκτός της μελέτης. Ε, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Ε, πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο παραγωγικό να υπάρχει μια αυξητική προσέγγιση και να πηγαίνουμε προς ε, ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ασύλου. Θα, υπάρχει ένα, θα υπάρχουν κοινά κέντρα ε, επεξεργασίας των αιτήσεων, ότι θα υπάρχει ένα νέο σύστημα ε, κατανομής της ευθύνης με αναθεώρηση του μηχανισμού του Δουβλίνου. Και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές. Και τώρα απαντάω στην κυρία Γιόμ. Δεν προτείνουμε νέο Δουβλίνο, προτείνουμε, λέμε ότι έχει φτάσει η στιγμή να εγκαταλείψουμε ε, το Δουβλίνο. Γνωρίζουμε ότι αυτό χρειάζεται πολιτική διαπραγμάτευση και μέχρι να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, και ε, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές δεν θα έπρεπε μέχρι τότε να είναι επιλογή ο εξαναγκασμός, γιατί αυτό αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο πνεύμα του συστήματος του Δουβλίνου προτείνουμε λοιπόν αυτήν την προσέγγιση. Για ποιο λόγο τώρα ε, το Δουβλίνο επαφίεται σε εσά ε, ως συνομοθέτη. Εν τω μεταξύ μπορείτε, εφόσον υπάρχει το Δουβλίνο, το εφαρμόζετε σωστά, βάσει των ε, υφισταμένων κανόνων. Και τώρα για την ερώτηση του κυρίου Λόπες Αγγιλάρ κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει μια ομάδα κρούσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ε, κάτι τέτοιο υπάρχει ήδη στη θεωρία τώρα. Κατά πόσο εφαρμόζεται, κατά πόσο ισχύει, αυτό είναι θέμα εντολής. Είναι το τι ζητούν τα κράτη-μέλη από το ΕΑΖΟ να κάνει και ε, ποια είναι η εποπτεία του Κοινοβουλίου σε σχέση με το τι κάνει το ΕΑΖΟ. Από την άλλη πιστεύουμε ότι το να τα αφήνουμε όλα στα χέρια όσων έχουν ευθύνη για την εφαρμογή των ε, νομικών κανόνων είναι επικίνδυνο. Οπότε θέλουμε να έχουμε λογοδοσία και διαφάνεια πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πιο πολυμερές σύστημα, το οποίο θα είναι πιο αξιόπιστο. Αν συμμετέχουν οι κυβερνητικέ οργανώσει, ε, η πατιαρμοστία του ΟΗΕ, ε, υπάρχουν περισσότερε πιθανότητες να υπάρχει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Τώρα για το ερώτημα που αφορούσε τις λύσεις. Οι προτάσεις, ε, οι εναλλακτικές για το Δουβλίνο υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά έγγραφα ε, και από το ΕΚΡΕ και από την ε, η, του ΟΗΕ. Σήμερα το απόγευμα νομίζω θα συζητήσετε αυτό το θέμα. Ε, όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει και το θέμα της επανεγκατάστασης. Όλα αυτά μπορούν να συσχετιστούν με την ε, συζήτηση για το Δουβλίνο. Υπάρχουν ήδη προτάσεις από κλίδα κατανομής, από ελεύθερη επιλογή, ε, να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των τούντων άσυλο ανάλογα με τους οικογενειακούς τους δεσμούς ή τη χώρα στην οποία θα θέλαν να καταλήξουν. όλα αυτά τα πράγματα βέβαια χρειάζονται νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι πέρα από αυτά που μπορούν να γίνουν βάσει του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως εντός του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου και κατά τη φάση της εφαρμογής των υπαρχουσών προδιαγραφών είναι όχι εξαναγκασμός. Μείωση του εξαναγκασμού τουλάχιστον αν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς τα, ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ως ε, οι ιδρυτικές ε, ε, αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως λέει και το άρθρο 8 είναι ήδη πάρα πολύ καλά. Καλό είναι λοιπόν να θεωρηθεί το Δουβλίνο ή να εγκαταληφθεί, αλλά ο, εφόσον δεν συμβαίνει αυτό ακόμα, τουλάχιστον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτού του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή. Για το πώς μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε. Πιλωτικά προγράμματα για την υποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων έχουν ήδη γίνει. Το ΕΑΣΟ το 2014 ε, έκανε πολλά πιλωτικά προγράμματα. Έγινε στη Βουλγαρία κάτι τέτοιο σε σχέση με την ε, εισρωή μεταναστών από τη Συρία ε, και μιλάω για τους όρους υποδοχής ε, και το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την υποστήριξη των μεταναστών στην Ιταλία. Όλα αυτά είναι ε, παραδείγματα ε, πρωτοβουλειών κοινών υποδοχής, κάτι το οποίο μπορεί να μας διδάξει και να μας βοηθήσει να βρούμε τη σωστή λύση για το μέλλον όμως ένα πλήρως, ολοκληρω, πλήρη ολοκληρωμένα κέντρα ασύλου πρέπει να ανταποκρίνονται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, πρέπει εκ των προτέρων να κατανέμεται η ευθύνη όχι μόνο σε σχέση με το ποιο κάνει τι, αλλά και πού θα γίνεται αυτό. Γιατί το κέντρο κάπου θα βρίσκεται εδαφικά, αλλά πρέπει το κράτος μέλος ε, που το φιλοξενεί να είναι πραγματικά ένας, ε, να είναι πραγματικά η υποδοχή με ό,τι σημαίνει αυτό αν ε, το κράτος μέλος ε, είναι υπεύθυνο πλέον για όλα όσα πρέπει να γίνονται στον τομέα του ασύλου, αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτό λοιπόν πρέπει εκ των προτέρων λαμβάνεται υπόψη. Μετά εκ των υστέρων θα πρέπει, αυτή στιγμή έχει ληφθεί η απόφαση, δεν πρέπει να μείνουν στα κέντρα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει κάπου να μεταφερθούν. Πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό και πάλι σημαίνει μεταφορές ατόμων. Και αν αυτές οι μεταφορές βασίζονται στο Δουβλίνο, εξακολουθεί να αποτελεί ο εξαναγκασμός τμήμα του συστήματος και εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι κρίσιμο το θέμα του εξαναγκασμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για το θέμα της πρόσβασης που θεωρείται το βασικό πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στη διαδικασία του ασύλου είναι το βασικό πρόβλημα. Οπότε, η κατανομή των ετούντων ε, έχει άμεση σχέση με το σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αυτό που κάνει το Δουβλίνο αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα, η θεώρηση των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθεί να είναι ότι το σύστημα είναι άδικο προς αυτούς. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί τελικά δεν στοιχειοθετούν αυτή τη θεώρηση. Οπότε η αποσύνδεση της κατανομής από το σημείο εισόδου, οποιαδήποτε κλίδα κατανομής θα αποφασιστεί, πρέπει να αποσυνδέει αυτά τα δύο πράγματα. Την κατανομή από την ευθύνη ε, της, ε, ε, του ελέγχου των συνόρων. Θέλει να επανέλθει, είχε ζητήσει, ήταν το μέλος που είχε αυτή την μελέτη. Παρακαλώ κύριε Νταγιόν, σύντομα. Και μετά να έχουμε καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Άκουσα πολλά σημεία. Τώρα που θα ήθελα να είναι αναλυτικά στην έκθεση και μια προσπάθεια να λύσουμε κάποια προβλήματα. Στην πρόταση δεν είπα. Δεν είχαμε πει ότι θέλουμε μεγάλη έκταση κέντρα και δεν συζητήσαμε για να δούμε τι εννοούμε. Πολλά φυσικά κάνατε. Πολύ το εξετάσατε. Αν έχετε στοιχεία και αν έχετε χρόνο, και δυνατότητα να εκπονήσετε ένα επιπλέον συμπληρωματικό υπόμνημα αλλά να μας αναφέρετε και λύσεις. Κοιτάξτε, είπατε ότι πρέπει να αναφερθούμε και στις πολιτικές πραγματικότητες. Ναι, μα εμείς είμαστε εδώ, είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε κυβερνήσεις και δεν μας ενδιαφέρει ο σχεδισμός δυνάμεων στο Συμβούλιο. Μπορούμε να σκεφτούμε ελεύθερα δεν πρέπει ε, μόνο μας κριτήριο να είναι η άποψη των κυβερνήσεων. Τώρα για τον ε, καταναγκασμό. Τι μας λέτε. Ότι η Ιρλανδία έχει καλό σύστημα ασύλου. Άρα καλύτερα να πάει κανείς εκεί για να ζητήσει άσυλο. Δηλαδή, εκεί που έχουμε τις καλύτερες καταστάσεις και τα υψηλότερα ποσοστά έγκρισης, θα πηγαίνουν οι περισσότεροι. Και αυτό είναι πολιτική πραγματικότητα. Όπως καταλαβαίνετε αυτό θα προκαλέσει επιδείνωση της λειτουργίας του συστήματος. Θέλουμε λοιπόν να εφαρμόζεται καλά το σύστημα παντού πριν πούμε ωραία τώρα πηγαίνετε όπου προτιμάτε. Ευχαριστώ Ντένις. Με συγχωρείτε γιατί ήθελε να επανέλθει. Θα πάρω την ε, Μαρή Λόριστον και μετά να κάνετε τα καταληκτικά σας σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα θαυμάσια μελέτη. Η ερώτησή μου και το σχόλιο. Βλέπω εδώ τους πίνακες όπου βλέπουμε πόσο διαφέρουν οι αριθμοί από την ίδια περιοχή από κράτος σε χώρα. Για παράδειγμα, από τις ίδιες χώρες προέλευσης, Σουηδία, Φινλανδία, πολύ διαφορετικότερες, ε, πολύ μεγάλη διαφορά, Ιταλία, Πορτογαλία, άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίσατε λοιπόν τη διαφορά συστημάτων και εφαρμογής του συστήματος για χώρες που από γενική άποψη είναι παρόμοιες. Μία λύση για να έχουμε ουσιαστική αλληλεγγύη θα μπορούσε να είναι μια πιο περιφερειακή προσέγγιση τα μεγαλύτερα αυτά κέντρα δεν θα πρέπει λοιπόν να αποφασίζονται στις Βρυξέλλες αλλά σε επίπεδο συνεργασίας χωρών παρομοίων παραδόσεων, πολιτισμού, νοοτροπίας. Για παράδειγμα στην ε, Βαλτική. Στη Σουηδία έχουμε 95, συγγνώμη, στην ε, Εστονία έχουμε 95 και στην Σουηδία έχουμε 54.000. Πολύ πιο εύκολο είναι να συμφωνήσουμε εμείς, μεταξύ μας εμείς οι δύο, παρά να συμφωνήσουν χώρες με πολύ διαφορετική προσέγγιση. Και επίσης ε, στις συνεντεύξεις που κάνατε δεν βλέπω να υπάρχει περιφερειακή προσέγγιση. Θα σας πρότεινα λοιπόν, και να και η ερώτησή μου, είναι δυνατόν να έχουμε μια πιο συγκριτική προσέγγιση και να συγκρίνουμε χώρες της ίδιας περιφέρειας. Ωραία, στις επόμενες συνεντεύξεις να συμπεριλάβετε και τη Βαλτική. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάγραμμα. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στα γραφεία μας. μόνο τέσσερις ή τρεις είναι οι χώρες στην ουσία που αντιμετωπίζουν σωστά. Λοιπόν, με αυτές τις ε, διακοπές τα τελικά σας σχόλια για να καταλήξουμε. Για αυτή την τελευταία ερώτηση, για την αλληλεγγύη. Να υπάρχει μια περιφερειακή προσέγγιση για να υπάρχει ουσιοδέστερη αλληλεγγύη. Ναι, γιατί όχι. Ναι, το επιτρέπει και η συνθήκη ήδη. Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης επιτρέπει και διμερή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, εάν το επιθυμούν. Υπάρχουν δυνατότητες ενισχυμένης συνεργασίας και διατάξεις που την προβλέπουν, αν κάποια κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Γιατί όχι. Αντί να έχουμε μια προσέγγιση είτε 28 είτε κανένας, που τελικά είναι λίγο άβολη. Ναι, μεν υπάρχει συναπόφαση, αλλά εντός του ΕΑΣΟ, εντός του συστήματος ασύλου, είναι δύσκολο να καταλήξουν όλα τα κράτη-μέλη. Για όλα τα υπόλοιπα, μία επιφύλαξη. Μερικές ερωτήσεις δεν εξετάστηκαν σε όσο βάθος θα θέλαμε γιατί αποφασίστηκε να λάβουμε την έκθεση τον Ιούλιο και έπρεπε να την παραδώσουμε το Σεπτέμβριο. Ε, σε δύο μήνες ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Ούτως ή άλλως, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη παραγγείλει μια σειρά από εκθέσεις για παράδειγμα για την εφαρμογή της ε, χρήσης ε, την εφαρμογή της αλληλεγγύης και τη δυνατότητα εκτός συνόρων να γίνεται αντιμετώπιση των ε, αιτήσεων. Δεν είχαμε δυνατότητα να δούμε τι έχει ε, γραφτεί για να έχουμε μία προσέγγιση σταδιακή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να επιτύχουμε κάποιες ε, επικοδομητικές λύσεις εντός του υπάρχοντος συστήματος, γιατί το Δουβλίνο 3 μόλις εγκριθεί, μόλις έχει εγκριθεί. Εάν λοιπόν δεν καταργηθεί αυτή η νομοθεσία, εάν δεν αναθεωρηθεί ριζικά, θεωρούμε παρόλα αυτά ότι μέχρι να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί από ένα Δουβλίνο 4 υπάρχουν πολλές δυνατότητε εφαρμογής τις οποίες μπορεί να επιτηρεί το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει συμμόρφωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ και τους τρεις συντάκτες. Ε, είπατε ότι ε, ε, συζητήσατε με ένα μέλος του Κοινοβουλίου, την κυρία Γκυγιό, μάλιστα, μεγάλη τιμή και ευθύνη. Σίλβια, δική σου είναι η έκθεση. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, συμμετοχή σας και παρουσίαση της έκθεσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η έκθεση αυτή για την περαιτέρω εργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, για το χρόνο σας. Στις 3 λοιπόν θα έρθει ο Αυστριακός Υπουργός για τα θέματα επανεκατάστασης.